Allora, possiamo... Ah, questo devo allora, ah, vabbè. allora intanto informo qual è l'ordine dei lavori così come è deciso ieri sera. σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που την αποφασίσαμε χθε το απόγευμα, τώρα πρέπει να κάνουμε τι ψηφοφορίε. Ναι. Για τις, ε, την πρακτική, τις πρακτικές λεπτομέρειες των εκλογών και μετά για την εντολή για τον προπολογισμό για τον τριμερή διάλογο. Τώρα, σε σχέση με τα, ε, θα σας ενημερώσω για το τι έγινε στους συντονιστές. Έπειτα έχουμε την έκθεση Fox για την έδρα του, των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Μετά έχουμε την έκθεση Γιαννάκου για το καθεστώ και τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ιδρυμάτων και πιο συγκεκριμένα για τον υποεξέλιξη τριμερή διάλογο. Και μετά έχουμε με βάση το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη το... Έχουμε λοιπόν τη δική μου έκθεση για την αξιολόγηση του προγράμματος της Στοκχόλμης καθώς και στη συνέχεια την έκθεση του κυρίου Τσαρκόφσκι για τις ψηφοφορίες και το περιεχόμενο των εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως στην ψηφοφορία για την ε, τροπολογία και τη συμβαστική 3 για την έκθεση του κυρίου Τσαρκόφσκι είναι υπέρ. Κατά. Εποχές. Ένας κατά και εγκρίνεται. Και αυτό σημαίνει πως καταπίπτουν έχουν λοιπόν καταπέσει η τροπολογίε 29 με 30 και περνάμε στην ψηφοφορία τη συμβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια. Και κοντράριο. Κατά. Αποχές. Τρεις αποχές και... Ε, τρεις κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν και η συμβαστική υπαριθμών 4 και τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 81 της κυρίας Μπελιέ, υπέρ. Και κοντράριο. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40 πρέπει να την ψηφίσουμε. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 λοιπόν, δε... όχι, τα μπέρδεψα. Τα μπέρδεψα, εντάξει, προχωράμε στην ε, τροπολογία 31, Σόλτς, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προχωράμε στην συμβιβαστική υπαρθμό 5. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως χρειάζεται να συμπεριληφθούν όλες οι πολιτικές, όλα τα πολιτικά κόμματα σε αυτή την παράγραφο. Μέχρι στιγμής απευθύνεται αποκλειστικά στα κράτη-μέλη, αλλά επίσης και τα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνη για να παρουσιαστούν στα ψηφοδέλτια ε, με τη μορφή που να επιλέγουν. Γι' αυτό πιστεύω πως θα ήταν καλό να πούμε καλούμε τα κρατημέλη και τα πολιτικά κόμματα να φροντίσουν ώστε τα ονόματα και όπου δει τα εμβλήματα ή τα σήματα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να εμφαίνονται στα ψηφοδέλτια. Οπότε ζητώ να συμπεριληφθούν αυτές οι τρεις λέξεις επιπλέον που λένε και τα πολιτικά κόμματα. Ο Γκουαλτιέρη. Ναι, ναι, ε, Συμφωνώ με την προφορική τροπολογία. Είναι κανείς αντίθετος στην προφορική, όχι. Ωραία. Με την προφορική τροπολογία ψηφίζουμε τη συμβαστική 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. 5 κατά καμιά αποχή. Τροπολογία 34 έχει καταπέσει, έχουν καταπέσει και οι άλλες και πάμε στην <clears throat> συμβιβαστική 6. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, καμία αποχή. Καταπίπτουν οι 41, 42, 43, 44, 46 και 42. Και πάμε στη 48 που πρέπει να ψηφιστεί, του κυρίου Χέφνερ. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Και κοντράριο. Κατά. Ε, Χρειάζεται να μετρήσουμε, παρακαλώ. Καλύτερα ηλεκτρονικά, ίσως. Έχετε τις κάρτες σας όμως. Εντάξει, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έχετε τις κάρτες. President, Πρόεδρε, δεν έχω εγώ την κάρτα ψηφοφορίας. Παρακαλώ, μετρήστε την ψήφο μου. Ούτε κι εγώ έχω την κάρτα. Υπομονή λοιπόν. α σηκώσουμε τα χέρια. Ε, ε, ε, Πρόεδρε, επειδή στο παρελθόν υπήρξαν προβλήματα σε αυτή την επιτροπή. Με την καταμέτρηση των ψήφων παρακαλώ να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία και μετά να μετρήσουμε χωριστά εκείνους που δεν έφεραν τις κάρτες τους. Νομίζω πως είναι σοφή η πρότασή σας, κύριε Ντάφ. Ψηφίζουμε μισό λεπτό τώρα γιατί ξέχασα που ήμασταν. Τροπολογία 47 Ντάφ. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Όχι. Όχι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Α, δεν λειτουργεί. Μα πρόεδρε τόσο δύσκολο να μετρήσουμε μέχρι το 12, να σηκώσουμε τα χεράκια μας να μας μετρήσετε. Μάλλον δεν ξέρετε και να χειριστείτε το μηχάνημα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και εγώ συμφωνώ Ας ε, είμαστε πιο ακριβείς. βάση περιπτώσει προσπαθούμε να φτιάξουμε το, το μηχάνημα. Άμα, άμα λειτουργήσει, μέχρι να λειτουργήσει, θα, θα συνεχίσουμε διανατάσσεως της χειρός. Ε, ε, Ο κύριος Νταφ, κοιτάξτε. Κάποιος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο εδώ, στην Επιτροπή μας στη γραμματεία και στη, διοίκηση που να ξέρει πώς να ανάψει το μηχάνημα και πώς να το ε, λειτουργήσει. Ναι, αλλά ειλικρινά. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά το γεγονό ότι ο επικεφαλή ε, τη Γραμματεία λείπει μα έχει δημιουργήσει κάποιε δυσκολίε. αν και κανονικά είναι κάτι είναι ένα θέμα ρουτίνα. εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να χάσουμε άλλο χρόνο για ένα θέμα το οποίο εύκολα μπορεί να λυθεί μέσω τη ψηφοφορία για να του χειρού και θα τα μετρήσουμε λοιπόν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, 47 ταφ είναι υπέρ παρακαλώ να σηκώσετε τα χέρια σας. Εγώ να σας μετρήσω.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 Τι λέτε εσεί 12. Ξανά μανά θα μετρήσω. Ποιοι είναι υπέρ. Πρώτα απ' όλα η αντιπρόεδρος. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 εντάξει 12 12 υπέρ κατά τώρα ποιοι είναι 12 12 12 9, 10, 11, 11. 11 quindi è approvato. 11 είναι κατά, άρα εγκρίνεται. Η 50 έχει καταπέσει. Το άρθρο 83 επίσης. Όχι 84 το ίδιο. Όχι, την 84 ψηφίζουμε, συγγνώμη. Μπελιέ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51. Έχει καταπέσει 49 όμως, ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά Πρέπει να μετρήσουμε υπέρ. 5, 6, 7, 8, 9. Contrari. Κατά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vabbè, respinto. Απορρίπτεται. 57. Favorevole. 57. Περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Ε, ναι, υπέρ. Θα μετρήσουμε για την 58. 7, 8, 9, 10, 11. 11 υπέρ, κατά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. È approvato. Όχι, δεν τα βρήκα. Ne ho contato 11 prima e, e, e Allora, siamo all'emendamento, scusate. Siamo eh, all'emendamento 58. 58, 58. Ο Νταφ. Κοιτάξτε. Μου φαίνεται ποιος πλέον δουλεύει το ηλεκτρονικό μηχάνημα. Παρακαλώ να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τη γραμματεία που άναψε το μηχάνημα. Λοιπόν, είστε όλοι έτοιμοι. Λάβετε θέσεις. Λοιπόν, είμαστε στην 57. 58, συγγνώμη, Σέφλιν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Άλλη μια φορά παρακαλώ. Okay. Okay. Okay, now. Ψηφίζουμε λοιπόν ξανά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Αποτελέσματα. Υπέρ 10 κατά 12. Εγώ θα ψηφίσει υπέρ, οπότε ψη... βάλτε και άλλη μια ψήφο. Υπάρχει άλλος που δεν ψήφισε, που δεν μπόρεσε μάλλον να ψηφίσει. Κύριε Γιαννάκου, δεν μπορέσατε να ψηφίσετε. 12-12 καταπίπτει πάντως τους ή άλλους γιατί έχουμε ισοπαλία. Απορρίπτεται λοιπόν.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 Όχι, τη Σέφελ δεν ψηφίσαμε, την 58, όχι την 85. Λοιπόν, απορρίπτεται 85, πάμε στην επόμενη 59, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Φτάσαμε στον συμβασμό 7, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν πάμε στις ε, τροπολογίες ε, συμβασμός 8, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται, που σημαίνει ότι καταπίπτουν οι 65, οι 66, Πάμε στην 67, παρακαλώ, ε, υπέρ, 67, κατά, αποχές απορρίπτεται. 68, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και φτάσαμε στην 69, υπέρ παρακαλώ, Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτήν. Συμφωνείτε όλοι. Πολύ ωραία λοιπόν. Ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 η 73 καταπίπτει το ίδιο ισχύει και για την 76 πάμε στην 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάσαμε τώρα στα ε, Υπάρχει μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ε, Κανεί τη διαφωνή. Υπέρ παρακαλώ. Στα εκτιμώντα, κατά αποχέ εγκρίνεται. Φτάσαμε στην τροπολογία 2. Ψηφίσαμε το εκτιμώντα 4. Πάμε στην ε, τροπολογία 2, στις αιτιολογικές σκέψεις, στην 4 ψηφίσαμε, πάμε τώρα στα επόμενα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 3 και οι 4 καταπίπτουν. ή 5 παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στο 6 υπέρ κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Έχω την εντύπωση ότι εγκρίνεται. Είμαστε στην 6 παρακαλώ. Α, volete fare il voto elettronico. Bene. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση, ε, την κάνουμε την επαλήθευση για το 6. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφορία. Έχουμε 13 υπέρ, 10 κατά, εγώ ε, θα ψήφιζα κατά. Εγκρίνεται. Η 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φτάσαμε στην 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά και ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ είμαστε στην 9 ψηφίζουμε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι να δούμε το αποτέλεσμα 8 υπέρ 15 ε, κατά άρα απορρίπτεται η 11 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, τροπολογία 10. Ψηφίζουμε παρακαλώ, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκανα ε, λάθος εκ παραδρομής, όπως λέμε. Ε, είπα το αντίθετο από αυτό που ήθελα να πω. Πάμε στην ε, τροπολογία, στο συμβασμό 2, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 16 τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Όχι, όχι, έχετε δίκιο. Προηγείται η 15 του κύριου Σόλτσε. Τροπολογία 15 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 14 καταπίπτει. Η... Μάλλον 14 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 του κυρίου Σόλτς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Βλέπετε το αποτέλεσμα 14 με 18, ακόμα και εγώ δεν θα άλλαζε τίποτα. Πάμε στο επόμενο, στο 19, Στο 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20, Ραντζέλ. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 15 με 7. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πολύ ωραία. Για την 22 λοιπόν, 22, ναι 22 Για την 22 δεν ψηφίζουμε, λέει ο Λοιπόν, ψηφίζουμε για την 22. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Εσείς λέτε 23. Α, ψηφίσαμε για την 22, συγγνώμη. Σωστά. Ε, ψηφίζουμε λοιπόν για την 23, την Σόπφλιν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά, έξι αποχές. possiamo 24. Για την 24 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25. Μισό λεπτό εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Dobbiamo votare? C'è un emendamento linguistico, è un problema di traduzione il 25. Uh, Κοιτάξτε, δεν, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για αυτήν. Ψηφίζουμε για την τελευταία τροπολογία, την 26, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν τούτου μπορούμε να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Ε, υπέρ παρακαλώ. Θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική θέλετε. Ναι, όχι. Ναι. Ωραία, ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ο κύριος Σόλτς. Κύριε Πρόεδρε, ξεχάσατε να ψηφίσετε, να ψηφίσουμε για την τροπολογία 43 και νομίζω ότι είναι σημαντική η τροπολογία αυτή. Για τη 43... Έχει πέρα καταπέσει. Page, page 3. Page 3. Non abbiamo votato, non is compatible with compromise 6 είναι ε, συμβατή με την έξι πρόεδρος. Μισό λεπτό, περιμένετε. Ε, δίκιο, δίκιο έχετε. Κατόπιν τούτου, πριν ψηφίσουμε για την τελική ψηφορία, να ψηφίσουμε για τη 43 του κ. Σόλτς υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και προσθέστε παρακαλώ και τη δική μου την ψήφο που είναι θετική. Πάρα πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν τώρα ε, στο... Εντάξει, συγχαίρουμε τον εισηγητή που πέρασε η έκθεση του και Περνάμε στην επόμενη έκθεση, την έκθεση του κυρίου Μέσα Σμιτ σχετικά με τον προπολογισμό του 2004, εντολή για τριμερή διάλογο. Τροπολογία 3, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5, υπέρ, Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 4. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την τροπολογία 5 λέει ο πρόεδρος. Την 4 την εγκρίναμε. 5 του ΝΤΑΦ. Υπέρ παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η δέκα ε, σε τμήματα ψηφίζουμε εδώ. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ε, πρέπει να κάνουμε έλεγχο παρακαλώ. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 10, ε, 3α. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και προστίθεται και η δική μου ψήφος που στην περίπτωση αυτή είναι καθοριστική γιατί είμαι αντίθετος, άρα απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 11. Χέφνερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 14 υπέρ 14 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πολύ ωραία. Για την τροπολογία 14 ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ας δούμε λιγάκι το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. 15, μάλλον 13 και 15 από κοινού. Καντίκου πρόεδρε, έχουν καταπέσει. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σας. Πολύ σωστά. Άρα έχουν καταπέσει. Πάμε στη 16 ε, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Για τη 17 δεν ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την τροπολογία 18. Έκλεισε η ψηφοφορία. Αποτέλεσμα παρακαλώ. Απορρίπτεται. Η 19. Τρακόφσκι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 του κύριου Νταφ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λάθος έκανα. Ψηφίσαμε για την τροπολογία Τρακόφσκι, ως εκ τούτου ε, καταπίπτει η τροπολογία Νταφ. Άρα δηλαδή λάβετε το υπόψη σας. Πάμε στην 21. Μπροτσμποχάτα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Νομίζω ότι καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. 21 μπροσάτα. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Και εδώ είναι καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά 22 Μπρτζοχομποχάτα υπέρ παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η ένα παρακαλώ υπέρ κατά νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι ίδια Απορρίπτεται απορρίφθηκε η 2 Τρτσκόφσκι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται που σημαίνει ότι τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ε, ψηφίσματος ηλεκτρονικά υπέρ παρακαλώ ψηφίζουμε μάλλον, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά έκλεισε η ψηφορία εγκρίνεται οριακά, προσθέστε και τη δική μου την ε, θετική ψήφο. Έχουμε δύο αποχές, με δύο αποχές λοιπόν. Πολύ ωραία. Και εδώ ε, τελειώσαμε με αυτή την ψηφοφορία. Ε, συγχαρητήρια και περνάμε στις ανακοινώσεις του Πρόεδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών. Allora, la riunione dei coordinatori ha esaminato in modo particolare. Εξέτασαν οι συντονιστέ λοιπόν το αίτημα 150 βουλευτών για επαλήθευση της Ε, συμμόρφωσης δύο κομμάτων με τις αξίες της Ένωσης. Η πρόταση που θα κάνουν οι συντονιστές στην Ολομέλεια της Επιτροπής μας είναι να γράψουμε μια επιστολή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν να λάβουμε κάποια απόφαση αυτή τη στιγμή, διότι δεν ε, υπάρχει αίτιο, δεν αιτιολογείται η μη συμμόρφωση. και στην επιστολή θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι βρίσκουμε ακατάλληλο, ότι δεν είναι δηλαδή δυνατό να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια της Επιτροπής μας, εφόσον δεν έχουμε στη διάθεσή μας μεγάλο γραπτό υλικό που υπάρχει στο Κοινοβούλιο, το οποίο εξέτασαν οι συνάδελφοι που θέλησαν να το κάνουν. Εξάλλου βρίσκεται σε εξέλιξη ο τριμερής διάλογος για το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων και σε κάθε περίπτωση αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα προηγούμενο το οποίο θα καθορίσει άσχημα τον ίδιο τον τριμερή διάλογο αρνητικά. Οπότε δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να αποφασίσουμε για να μας δώσει ενδεχομένως περαιτέρω οδηγίες. Επίσης αποφασίσαμε να αλλάξουμε τον τίτλο της έκθεσης ε, που λέει ε, τέσσερα χρόνια μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι να κατάλληλος αυτός ο τίτλος γιατί κατά κάποιο τρόπο ε, αντιτίθεται στην έκθεση Γκουαλτιέρη και Λαμασούρ και έτσι σε λίγο ο κύριος Σταρκόφσκι σε λίγες μέρες καθώς είναι το ΕΛΚ που έχει αναλάβει αυτή την έκθεση και ο Ρανζέλ νομίζω θα μας δώσει έναν διαφορετικό και πιο συγκεκριμένο τίτλο για την έκθεση αυτή. Lo detto così, no? Oh. Eh, Va bene. Poi il, per quanto riguarda altre relazioni di iniziativa, io ho... Όσον αφορά άλλε εκθέσει πρωτοβουλία, ε, Ζήτησα εγώ μια έκθεση πρωτοβουλία για τι σχέσει ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ζητήσουμε αυτή την έγκριση γιατί πετύχαμε έγκριση για πέντε εκθέσεις πρωτοβουλίας. Ωστόσο, πρέπει να επιμείνουμε στην διάσκεψη των Προέδρων για να γνωρίζουμε αν όλες αυτές οι εκθέσεις πρωτοβουλίας που ήδη έχουμε ζητήσει εγκρίνονται ή όχι. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την από την ε, πόση ενός εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτό δεν γίνεται, θα το ζητήσουμε ως χωριστή ε, έκθεση. Επίσης ενημερώνουμε την Επιτροπή πω το Συμβούλιο θα διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο προς έγκριση το σχέδιο απόφαση που ορίζει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιση των εκλογών του 2014 και επειδή αυτό φαίνεται να επίκειται και δεν υπάρχει πολλή χρόνος προτείνεται να διοργανωθεί μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για την Δευτέρα 10 Ιουνίου στο Στρασβούργο, ώστε να μπορέσουμε σύντομα να εγκρίνουμε αυτό το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου. Οι συνεισηγητές για αυτή την έκθεση του, του Κοινοβουλίου είναι ο Γκουαλτιέρη και ο Ταρκόφσκι, ο οποίος ε, θα πρέπει να μας επιβεβαιώσει ότι θα είναι εκείνο. Στην έκτα της συνεδρίας του Στρασβουργού θα, μπορούσε επίσης να ακούσουμε, θα μπορούσαμε επίσης να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εύκοβιτς, ο οποίος, ως ήθιστε, έχει προσκληθεί για να κάνουμε τον ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο για τις εξελίξεις και την ανάπτυξη της δικής μας Επιτροπής τα τελευταία πέντε χρόνια. Έπειτα, η αντιπροσωπεία που θα πάει στο Λονδίνο 19 και 20 Ιουνίου, η αντιπροσωπεία εκτός από τον Πρόεδρο θα πρέπει να αποτελείται από δύο μέλη του ΕΛΚ, ε, δύο σοσιαλιστές και έναν για το κάθε μία από τις άλλες ομάδες. Μέχρι τώρα όμως, πέρα από τον Πρόεδρο, είναι η κυρία Λεγκρίπη, Σέφλινγκ, Ταρκόφσκι, Γουαλτιέρη, Ιλκ, Χέφνερ και Σόλτς. Υπάρχει ένα αίτημα... Όχι, οι συνάδελφοι από το Ηνωμένο Βασίλειο Ντάφ και Άγνιου θα συμμετέχουν εκτός ποσόστοσης όπως ήθιστε. Το ΕΛΚ έχει παρουσιάσει τρία μελέτη για δύο, αλλά αυτό το είχαμε συμφωνήσει. Και έπειτα υπάρχει και περαιτέρω ετοιμα ακόμα δύο μελών. Μάξιμο όμως έναν ακόμα θα αφήσει η ε, διάσκεψη των πρόεδρων να έρθει. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από πλευρά της Επιτροπής, Αυτά είναι τα όσα συμφώνησαν οι συντονιστέ. Αν το εγκρίνει η διάσκεψη του Πρόεδρου, ο συνάδελφο Χέλμαρ Μπρόκα θα συμμετέχει και κινούσε στην αντιπροσωπεία στο Λονδίνο. Αυτέ είναι οι ανακοινώσει και περνάμε στο άλλο σημείο τη ημερήσια διάταξη, το επόμενο που αφορά. Che riguarda e τις εκθέσεις Φόξ και Χέφνερ. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω από την Αντιπρόεδρο Κουρμάη να αναλάβει σε αυτή τη φάση την Προεδρία. Διότι εγώ χρειάζεται να λείψω για ένα λεπτό. Okay, so, uh, thank you very much, dear Σας ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ήμουν ε, τυχερή που προείδρευσα χτες στην ε, πολύ πετυχημένη δημόσια κρόση και είμαι πολύ ε, ευτυχής και ευχαριστώ τους συναδέλφους που το διοργάνωσαν. Ήταν εξαιρετικοί οι τέσσερις εμπειρογνώμονες που ήταν εδώ εχθές. Θα ήθελα να ρωτήσω απλά ποιος θέλει να ξεκινήσει, να, μιλήσει, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ναι, ο κύριος Φόξ που είναι ο Παρακαλώ. Κυρία Κύριε Πρόεδρε, Καταρχήν θέλω να σου πω, ζητώ συγγνώμη, ότι 11 και 20 πρέπει να φύγω και ήδη έχουμε καθυστερήσει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα μιλήσω μόνο για λίγο και μετά ο Γκέραλτ θα ολοκληρώσει τη συζήτηση. Όπως πολύ σωστά είπατε, εχθές είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Συζητήσαμε για το τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου, κυρίως για το δικαίωμά του της ε, αυτοοργάνωσης. Έχουμε λοιπόν ένα έγγραφο εργασίας που αφορά ε, στην έδρα των ευρωπαϊκών θεσμών. Το έγγραφο αυτό προηγείται του ε, σχεδίου το οποίο σύντομα θα καταθέσω στους συναδέλφους. Θα γνωρίζετε ότι η δική μας έκθεση πρωτοβουλίας είναι πολύ περιορισμένη, τουλάχιστον όσον αφορά το την έκτασή τη. Ε, γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτό το έγγραφο εργασίας για να εξηγήσουμε λιγάκι το σκεπτικό της έκθεσής μας. Μπορείτε να βρείτε το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις ε, έδρες των ευρωπαϊκών θεσμών. Παρουσιάζουμε τις ιστορικές εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ε, αναφέρουμε ε, το ότι κατά την άποψή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη αυτονομία όσον αφορά τις έδρες της και το χρονοδιάγραμμα εργασιών κατόπιν αναλύουμε τις ε, περιβαλλοντικές ε, και άλλες επιπτώσεις των ισχυουσών ρυθμίσεων. Και καταλήγουμε με αυτό που κατά την άποψή μας είναι ο χάρτης πορείας προς την κατεύθυνση της αλλαγής των ε, συνθήκων. Νομίζω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει και αυτό το έχει δείξει τα τελευταία δύο χρόνια μέσω διαφόρων ψηφοφοριών ότι επιθυμούμε όλες μας οι συνεδριάσεις να λαμβάνουν χώρα σε μία και μόνο έδρα. Ε, βέβαια, ε, διάφορα μέλη έχουν τους δικούς τους λόγους ο καθένας ε, για να στρίξουν αυτή την άποψη. Για κάποιους είναι τα χρήματα των φορολογουμένων, για άλλους το διοξίδιο του άνθρακα και για άλλους πάλι διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει την δυνατότητα να αυτοοργανώνεται. Αυτό όμως που είναι απόλυτα σαφές είναι ότι διαγράφεται πλέον πλειοψηφία ανάμεσα στους βουλευτές ότι όλες οι συνεδριάσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε μία και μόνο έδρα. Βεβαίως ο Γκέραλτ και εγώ δεν λέμε σε ποια έδρα, δεν, ε, δεν εκφράζουμε την προτίμησή μας γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος της έκθεσης. Δεν λέμε, δεν είναι δική μας δουλειά να πούμε ότι όλες οι συνεδριάσεις να λαμβάνουν χώρα στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού. Εκείνο το οποίο εμείς λέμε είναι ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει για το θέμα της έδρας και το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει πού θα λαμβάνουν χώρα οι συνεδριάσεις. Σε αυτό λοιπόν το έγγραφο εργασίας έχετε το σκεπτικό της ε, πρότασής μας ε, και έχετε επίσης και την ε, πρόταση και τη συστάση. Αυτές μάλλον θα τις έχετε συντομότατα. Αυτά είχα να σας πω κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που είμαι αναγκασμένη να φύγω σε 20 περίπου λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνεισηγητής Γκέραλτ Χέφνερ έχει το λόγο. Θα παρέμβω στη συζήτηση και θα μιλήσω στο τέλος. Ε, για εισαγωγή νομίζω αυτά αρκούν. Και ε, για τον Άσλι Φόξ και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα να ακούσουμε πλέον τα σχόλια των συναδέλφων για το έγγραφο εργασίας μας και να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για έγγραφο εργασίας έτσι δεν είναι το σχέδιο έκθεσης αυτό. Ε, θα το επεξεργαστούμε αυτό το σχέδιο υπό το φως της σημερινής συζήτησης. Γι' αυτό περιμένουμε να ακούσουμε τα δικά σας σχόλια για να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Και η χθεσινή συζήτηση πιστεύω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ. Ε, για... Ο κύριος Ρούτσας και ο συγητής, θέλει το λόγο. Α, πρώτα ο κύριος Ρομπέρτο, συντονιστή συντονιστής των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Δυστυχώ πρέπει να φύγω, να πάω στο Προεδρείο τη ομάδας μου, γι' αυτό και ο συζητητής μα θα παρα... μάλλον θα σας εξηγήσει πιο λεπτομερώς ε, ε, τις θέσεις μας. Μερικά σχόλια για το έγγραφο εργασίας θέλω να κάνω. Ε, από τη σκοπιά κάποιου που είναι ακρεφνής υποστηρικτής της μίας έδρας, αλλά έχει κάποιες επιφυλάξεις για τη γραμμή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, ο βασικός μας ισχυρισμός θα πρέπει να είναι ότι το Κοινοβούλιο και μόνο το Κοινοβούλιο αποφασίζει για την έδρα του. Ε, και το θέμα αυτό είναι συνταγματικής φύσεως. Και σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε χθες το άρθρο 341 της συνθήκης δεν ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 10 ε, της συνθήκης διότι ε, τα κράτη-μέλη ε, αλλά και οι πολίτες ορίζουν τη νομιμότητα τη Δημοκρατική Ενώση Κοινοβουλίου. Προτιμώ να θεώρηση της συνθήκης που να καθορίζει διαφορετικά την έδρα. Θα τα εξηγήσει αυτά ο κύριος Δρούτσας. Να κάνω όμως ένα γενικό σχόλιο της συνταγματικής φύσεως. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να συγχέουμε ε, το τρόπο εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας με το θέμα της έδρας των θεσμικών οργάνων. Ε, είναι αντιπαραγωγικό ενδεχομένως αυτό και επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να φαίνεται πιο εύκολο να πούμε ότι δεν επιλέγουμε μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου. Απλώς θέλουμε να είμαστε εμείς εκείνοι που θα αποφασίζουμε. Αλλά το να ζητάς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αφήσει στα χέρια του Κοινοβουλίου αυτό το θέμα, που είναι και πολύ χαμηλό το κατόφλι κατά τα άλλα της ειδικής πλειοψηφία της ενισχυμένης που χρειάζεται, Δηλαδή κατά πλειοψηφία θα ε, αποφασίσουμε για το, σε ποια πόλη θα είμαστε Αφήστε που μπορούμε να αποφασίσουμε και ένα τελείως διαφορετικό μέρος, πιο ζεστό, πιο ηλιόλουστο κτλ. Ε, ε το θέμα αυτό ε, είναι θέμα συνθήκων. Σε αυτό το συνταγματικό επίπεδο θα πρέπει να συζητηθεί. Και μάλιστα μαζί με τους εκπροσώπους των πολιτών αλλά και των κρατών μελών. Είναι διπλή εκπροσώπηση. Και σύμφωνα με την άποψή μου θα πρέπει να είναι πιο ορθολογική η οργάνωση. Οι δύο βραχίονες ε, της νομοθετικής εξουσίας θα πρέπει να συναποφασίζουν ε, άρα και να εδρεύουν ε, στην ίδια πόλη. Αυτό είναι λίγο το στοιχείο που δεν με πείθει η συνταγματική η στρατηγική. Και με ποιο τρόπο μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι έγγραφο εργασία. Γι' αυτό και η χθεσινή ακρόαση που κάναμε ε, μας διαφωτίζει λίγο περισσότερο για να είμαστε και πιο επαγγελματικοί στην προσέγγιση μα. Να σα πω ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο για να ε, βεβαιωθούμε ότι σας έχω όλους δει και σημειώσει. Λεγκρίπ Δρούτσας, Βίλαντ, άλλος κανείς, παρακαλώ, Νταφ Μπρόνς, άλλος, αυτή. Λοιπόν, η Αντιπρόεδρος η κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να κάνω μερικά σχόλια για το έγγραφο εργασίας που μας παρουσιάζεται σήμερα. Και χτες το απόγευμα μίλησα και εξέφρασα ε, την έκπληξή μου ως προς την επικεφαλίδα, τον τίτλο της πρόσκλησης στην ακρόαση, που ε, ελαφρά την καρδία, αναμείγνυε τον τόπο εργασίας, την έδρα. Ήταν πραγματικά πολύ μονόπλευρη και μεροληπτική αυτή η πρόσκληση. Και ε, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον τίτλο της έκθεσης πρωτοβουλίας, όπως αποφασίστηκε στην Επιτροπή και στη συνέχεια εγκρίθηκε στο Προεδρείο, και στη συνέχεια το περιεχόμενο που προσέλαβε. Δηλαδή σε τέτοιο βαθμό που οι ίδιοι οι συνεισηγητές μας λέγουν ότι είναι έκθεση για την έδρα ε, των θεσμικών οργάνων γενικώ, αλλά ας επικεντρωθούμε στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, ας μην είμαστε γνωρίζουμε πολύ καλά το πλαίσιο στο οποίο περιγράφονται οι εργασίες μας, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω για να ακουστεί. Διότι κατά την άποψή μου το θέμα των εδρών όλων λέει, των θεσμικών οργάνων της Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με άλλα ζητήματα και πολιτικά και νομικά. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε ε, το θέμα της έδρας ενός και μόνου θεσμικού οργάνου από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και οργανισμούς. Αυτό για τον τύπο ε, ως σχόλιο. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Πολλά είναι εκείνα που δεν μου αρέσουν σε αυτό το έγγραφο εργασίας και το επαναλαμβάνω. Το κείμενο που μας ε, κατατίθεται σήμερα ε, έτσι πάρα πολύ αβασάνιστα συγχαίει διάφορα πράγματα και προσθέτει σύγχυση ανάμεσα σε τόπο εργασίας και έδρα. Ε, αναμειγνύονται αυτές οι έννοιες, υπάρχουν κάποια σφάλματα και εκτιμήσεις που δεν μπορούμε να δεχτούμε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, να διασκεδαστεί η σύγχυση αυτή. Όλοι γνωρίζετε ότι μία είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα πρέπει να γράφουμε ε, πράγματα σύμφωνα με τις συνθήκες και να σεβόμαστε τις συνθήκες στις διατυπώσεις μας. Επίσης, στην παράγραφο 3, ιστορικές εξελίξεις, νομίζω υπάρχουν κάποιες ε, ελλείψεις. Ε, έχουμε λησμονήσει ότι στο Εδιμβούργο δεν αποφασίστηκε μόνο το θέμα αυτό της ε, εκ νέου διατράνωσης της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβουρού. Υπήρχε και άλλη απόφαση τότε στο Εδιμβούργο, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εγκατασταθεί κάπου στη Γερμανία και άλλες έδρες δηλαδή διανεμήθηκαν και άλλοι οργανισμοί ε, σε άλλες χώρες. Δεν ήταν μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό επανέρχομαι ε, στο προηγούμενο ότι είναι όλα αυτά πάρα πολύ μπερδεμένα μεταξύ τους και δεν θα πρέπει να λησμονούμε τις ιστορικές εξελίξεις όταν κάνουμε μια τέτοια ιστορική αναδρομή. Στην παράγραφο 3 επαναλαμβάνω του εγγράφου εργασίας που μας έχει υποβληθεί. Και τον Απρίλιο του 1991 επίσης είχε ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και οι βουλευτές ε, υπερψήφισαν. Αυτό που τελικά ε, ονομάστηκε ε, Συμβασμός Πέτερς. Όπου και πάλι είπαμε διατρονώθηκε ε, το θέμα της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίστηκε στο Στρασβούργο. Λοιπόν, μια που είμαστε εδώ Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και έχουμε και ολόκληρη έκθεση πρωτοβουλίας για το δικαίωμα του Κοινοβουλίου στην αυτοοργάνωση. Και μάλιστα το τραβάμε τόσο πολύ μέχρι που να μπορεί να επιλέγει το κοινοβούλιο την έδρα του. Πρέπει να πω ότι διαφωνώ και έχουμε και μια δυσφορία σε σχέση με αυτό ε, και ε, όλη την παράγραφο 5 που είναι εκτός θέματος, εν πάση περιπτώσει είναι εκτός πεδίου αρμοδιοτήτων της δική μας Επιτροπής. Παράγραφος 5 που λέει οικονομικά, περιβαλλοντικά, οργανωτικά στοιχεία και επιμελητία. και αρχίζει εδώ με διάφορα αριθμητικά στοιχεία να υπολογίζει και στοιχεία που είναι τελείως εκτός αρμοδιοτήτων. Αφήστε που θα τα αντικρούσω και θα τα καταρρύψω ορισμένα. Τι δουλειά έχει αυτό σε μια νομική συζήτηση και συνταγματική για τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το κατά πόσο ε, είναι θεμητό να ορίζει τον τόπο στον οποίο εδρεύει και πώς θα οργανώνεται και πώς θα λειτουργεί. Μιλάνε εδώ για ε, αεροπλάνα, τρένα, ξενοδοχεία. Το μόνο που έλειπε να μας πούνε είναι καθαρά τα πεζοδρόμια ή τα ταξί. Τι δουλειά έχουν αυτά σε ένα έγγραφο, έστω και έγγραφο εργασία. Ξέρω ότι δεν είναι σχέδιο έκθεση, ε, αλλά θα ακολουθήσει η έκθεση πρωτοβουλία. Τι δουλειά έχει αυτή η παράγραφο σε ένα τέτοιο έγγραφο τη Συνταγματική Επιτροπή. Έλεω, συνάδελφοι. Ε, αν έλθουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο συζήτησης και να μην βγαίνουμε από το πεδίο που μας αναλογεί. Και επίσης τα στοιχεία τα αριθμητικά εγώ τα αμφισβητώ το εγγράφου εργασία στη παράγραφο 5. Έχουν βγει κατευθείαν από έγγραφα προπαγάνδας ε, εκείνων που προωθούν το one single seat ε, που θέλουν να έρθουν άλλα στις Βρυξέλλες. Και αυτά τα στοιχεία εμεί τα αμφισβητούμε και όχι μόνο εγώ, είμαστε πολλοί, είναι απαρχιωμένα, δεν ισχύουν ε, και δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν απαντά, ας πούμε, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για την απαλλαγή, υπάρχουν επίσημα στοιχεία που δίδει ο Γενικός Γραμματέας ε, του Κοινοβουλίου. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτά. Ας πούμε, το κόστος που υπολογίζεται και πάλι βάσει των επισήμων στοιχείων έτσι του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου ε, για τους πολλούς τόπους εργασίας είναι 51,5 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ διαφορετικό ως τάξη μεγέθους από αυτό που αναφέρεται εδώ στην έκθεση. Επίσης, ε, το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα. Επίσημα στοιχεία, επαναλαμβάνω, του Γενικού Γραμματέα είναι πιο κοντά στις 4.199 τόνους και πολύ λιγότερο σε αυτά που αναφέρετε εσείς. Λοιπόν, αυτή η παράγραφος 5 είναι απόπειρα διακρίσεων και ε, κάποια στοιχεία κατά προσέγγιση, όχι ακριβή και πιστεύω ότι είναι τελείως περιττό και άσκοπο να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις και μάλιστα με στοιχεία πάρα πολύ αμφισβητούμενα, αμφισβητήσιμα και καλό θα ήταν να παραμένουμε σε επιχειρήματα που αφορούν τη δική μας επιτροπή και είναι λίγο έτσι, ανωτέρου επίπεδου. Ε, ακούστηκαν πολλά εχθές κατά τη διάρκεια τη κρόασης, πολύ διαφωτιστικά όσο και ενδιαφέροντα. Είχαμε και πολλούς εμπειρογνώμονε. Σημειώνω ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επανειλημμένα δις ε, ξεκαθάρισε τα πράγματα και επεφάνθη ότι δεν υπάρχει περιορισμός της εξουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ε, στο δικαίωμα αυτοοργάνωσης ή αυτοτελούς λειτουργίας διότι οι συνθήκες ορίζουν την έδρα του. Λοιπόν, δύο φορέ απεφάνθη από αυτό το δικαστήριο ότι δεν περιορίζονται εξουσίε και αρμοδιότητε από αυτό το θέμα και επίση από τη χθεσινή ακρόαση τη βγήκε, τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ και αντιλαμβάνομαι του εμπειρογνώμονε, ότι το θέμα τη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί αυτό μα απασχολεί και όχι των άλλων θεσμικών οργάνων από ό,τι φαίνεται, ε, είναι κάτι που έχει οριστεί σε ένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών μελών και των εκπροσώπων των πολιτών. Είπαμε υπάρχει αυτή η διπλή πολιτική νομιμότητα ε, και δημοκρατική νομιμότητα στην Ευρώπη. Αυτά δεν θα πω κι άλλο τώρα στο παρόν στάδιο, αλλά νομίζω χρειάζεται κάποια επανεξισορρόπηση το κείμενο για να είναι λίγο πιο αναβαθμισμένο και να αναφέρει και πραγματικά στοιχεία και όχι κάποιες ε, αμφισβητήσιμες και αμφισβητούμενες ε, υποθετικές παραδοχές. Αυτά. Ας επανέλθουμε επίσης στο συνταγματικό πεδίο και ας αφήσουμε αυτή την παράγραφο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλους πέντε ομιλητές, συν ε, των Παρακαλώ, εκαστος τρία λεπτά ε, και μετά πέντε λεπτά για τον κύριο Χέφνερ. Επόμενος, είναι ο κύριος Δρούτσας, παρακαλώ, και ο δισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω τα τρία λεπτά. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές ε, για το έγγραφο εργασίας και γενικότερα για τη δουλειά τους. Τους ευχαριστώ για το πνεύμα συνεργασίας και επίσης ε, διότι ευθύς εξ αρχής ε, προσπάθησαν να διατηρήσουν την επαφή με όλους μας και να εκφράσουν τις ε, απόψεις τους. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και πιστεύω ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση ανάμεσα στους συναδέλφους και τις πολιτικές ομάδες. Είχαμε τη χθεσινή ακρόαση Ακούσαμε τους ε, εμπειρογνώμονές μας. Εγώ ε, κατάλαβα τουλάχιστον ότι πρόκειται για ένα αμυγός ε, πολιτικό θέμα, μια ξεκάθαρη πολιτική απόφαση. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι εγώ δέχομαι την προσέγγιση των συνεισηγητών, δηλαδή να εξετάσουμε το θέμα κάτω από διαφορετικό πρίσμα, ότι θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα ως Κοινοβούλιο να αποφασίζουμε μόνοι μας, να οργανώνουμε μόνοι μας το ε, χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας και να ορίζουμε μόνοι μας την έδρα όπου θα συνεδριάζουμε. Θέλω μόνο να πω ότι υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτα απ' όλα, το αποτέλεσμα δεν θα είναι διαφορετικό ε, αν δεχτούμε αυτή την προσέγγιση ή την παραδοσιακή που λέει ε, επί το θέμα της έντρας ε, να αποφασίσουμε αν θα είναι Στρασβούργο ή Βρυξέλλες. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια αλλαγή των συνθήκων. Είναι απαραίτητο να πράξει και μια διακυβερνητική συνέλευση. Όπως είπε και ο κύριος Γκουαλτιέρη, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το θέμα. Δηλαδή, κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μπορεί να αποφασίσει μόνο του. Πρέπει να το κάνουμε αυτό ή μήπως ε, αυτά όλα θα πρέπει να ρυθμιστούν από τις συνθήκες χτες από την ακρόση εγώ δεν κατέληξα κάπου συγκεκριμένα. Γι' αυτό λοιπόν ε, παρακαλώ τους ε, συνεισηγητές να το δουν το θέμα προσεκτικότερα και να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα επ' αυτού του θέματος. Όσον αφορά τώρα στο έγγραφο εργασίας θα μου επιτρέψετε κυρία Αντιπρόεδρε να έχω διαφορετική άποψη από εσάς. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσέγγιση και επίση και από τον τρόπο με τον οποίο συντάχθηκε το έγγραφο εργασίας. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν και λεπτομέρειες, να υπάρχουν ονόματα, να υπάρχουν αριθμοί, γιατί πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επίμαχο θέμα, άρα δηλαδή τα επιχειρήματα είναι σημαντικά. Και επίσης είναι και απαραίτητο ο Ευρωπαίος πολίτης να έχει στη διάθεσή του τεκμηριωμένες πληροφορίες η δική μας έκθεση μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως έχετε δίκιο ότι αν υπάρχουν διαφωνίες επί των αριθμών, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικό από αυτού, αν αμφίβολα και εδώ απευθύνομαι στους συνεισηγητές, παρακαλώ ε, δώστε μας τεκμηριωμένες πληροφορίες ή τουλάχιστον υπάρχει μια δυνατότητα επαλήθευσης των ε, υποβαλόμενων στοιχείων. Πάντως σαφώς και είμαι υπέρ αυτού που προτείνουν οι συνεισηγητές. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στην έκθεσή μας. Και δύο δευτερευούσεις φύσεως ε, θέματα σχετικά με την έκθεση. Έχουμε την επικεφαλίδα που λέει έκθεση για τις έδρες των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση όμως γίνεται αναφορά μόνο στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνω βέβαια όλο το σκεπτικό, αλλά εγώ προτείνω να προσαρμόσουμε και την επικεφαλίδα της έκθεσής μας, γιατί για μένα αποτελεί σαφή αντίφαση το ότι στην επικεφαλίδα γίνεται λόγος για τις έδρες όλων των ευρωπαϊκών θεσμών και μετά γίνεται λόγος μόνο για την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν να το δούμε το θέμα αυτό. Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει ή είναι απαραίτητο να υπάρξει και κάποια άλλη ε, διευκρίνηση, καθότι το έγγραφο εργασίας μιλάει για μια κανονική διαδικασία με βάση το άρθρο 48 και στην επόμενη παράγραφο στο τμήμα 6 του εγγράφου εργασίας λίγο πολύ γίνεται λόγο σε μια, για μια απλουστευμένη διαδικασία. Επίσης ε, Αναφέρεται ότι υπάρχουν κάποια παραδείγματα του Ευρωπαϊκού ε, Μηχανισμού Σταθεροποίησης ότι αυτός ας πούμε δεν έχει καμία σχέση με τη συνθήκη. Νομίζω αυτό πρέπει να το αλλάξουμε λιγάκι και πρέπει να στοχεύουμε στο να έχουμε μία ε, καθαρή γλώσσα κυρίως όταν πρόκειται για νομικής φύσεως θέματα. Και το τελευταίο κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου το υπενθυμίσατε λέει ο θεωρώ ότι είναι χρήσιμο στην έκθεση να αναφέρεται και το θέμα των προτάσεων ή σκέψεων για την εναλλακτική χρήση του Στρασβούργου. Αναφέρθηκαν τόσες πολλές ιδέες, ας πούμε από το σημαντικότερο να συνεδριάζει στο Στρασβούργο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, και με αυτόν τον τρόπο να διατηρείται η συμβολική και ιστορική αξία του Στρασβουργού ή στο Στρασβούργο να συνεδριάζει η Επιτροπή των Περιφερειών. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό ε, να αναφερόμαστε και στο ποιες θα μπορούσαν να είναι οι εναλλακτικέ λύσεις για το Στρασβούργο. Ευχαριστώ είστε μεν σκιώδη, αλλά σα ζήτησα ευγενικά να αφήσετε και λίγο χρόνο στον εισηγητή μα, τον κύριο Χέφνερ. Αντιπρόεδρος κύριο Βίλαντ είναι ο επόμενος ομιλητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κατανοώ το μέλημά σας, αλλά σε κάποια σημεία του εγγράφου ε, βλέπω ε, ότι προσπαθούν να μας περάσουν διάφορα πράγματα. Ε, υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις του τύπου κατόπιν πιέσεως της Γαλλίας που μου φαίνονται άσκοπες. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, τελικά μόνο θα διαπληκτιστούμε. Και κάποιοι φανατικοί των αριθμών που πάντα μιλούν για το κόστος δεν μπορούν να μας απαντήσουν γιατί τόσο καιρό όταν είμαστε στο Στρασβούργο αφού πηγαίνουμε στο Στρασβούργο έτσι και αλλιώς γιατί να μην συνεδριάζουμε πέντε μέρες και πολύ γεμάτες και αποτελεσματικές και όχι τέσσερις. Αυτοί που προφασίζονται πάντα το κόστος θα πρέπει να διαρωτηθούν και ίδιοι κάποια πράγματα. Και ένα τελευταίο. Στην όλη συζήτηση εγώ τουλάχιστον θα προσέξω πάρα πολύ πού βρίσκονται οι αντίπαλοι του Κοινοβουλίου και τι λένε για την έδρα και τι λένε για την έδρα οι φίλοι του Κοινοβουλίου. Διότι ε, πιστεύω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ανίερες συμμαχίες. Ειδικά αυτοί που ενδιαφέρονται για την αυτοοργάνωση, για την έδρα, δεν είναι πρόθυμοι στο Κοινοβούλιο να δώσουν ε, ούτε ίχνος περισσότερων εξουσιών και δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Εγώ δεν θα πεθάνω, υποστηρίζω το Στρασβούργο. Αλλά ανέκαθεν έλεγα ότι αν είχα δικαίωμα ε, το Κοινοβούλιο να αυτοοργανώνεται, να το κάνουμε και να αποφασίζει τελικά για θέματα έδρας και η Ολομέλεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί εκεί μπαίνουν και ζητήματα καθεστώτος, ασυλίας και πολλά άλλα όπου θα πρέπει να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να αποφασίζει, επιτρέπεται μόνο του το Κοινοβούλιο, ενώ κάποια άλλα μπαίνουν σε μια συντεταγμένη συναπόφαση, όπου και το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να μπορεί να κρυφτεί πίσω από την ομοφωνία. Γι' αυτό επίμεινα η ακρόαση να γίνει υπό τον τίτλο υπό τον οποίο έγινε. Το θέμα της έδρας ε, το θεωρώ πολύ μονοδιάστατο για να αναχθεί σε αυτό και να περιοριστεί. Θέλω μια συνολική προσέγγιση. Και μετά να έχετε και την ψήφο μου. Εάν είναι προφάσεις μόνο μαρτίες για να καρατομηθεί το Στρασβούργο, δεν θα σας δώσω ε, την ε, ψήφο μου και μάλιστα υπό καμία περίπτωση. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω όλους να έχουμε μια προσέγγιση και να επιλέξουμε πιο συνολική. Και κατά τα άλλα πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πολύ χρόνο αν αυτοί που δεν τηρούν το χρόνο αρχίζουν την ομιλία τους λέγοντας ότι θα τον τηρήσουν. Ευχαριστώ ο κύριος Νταφ και μετά ο κύριος Μπρός. Um, uh, Συμφωνώ πως ε, χρειάζεται να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε την περιπλοκότητα και την ε, λεπτότητα του θέματος και νομίζω, όπως είπε και η Κωνσταντς Λεγκρίπα, ότι κάποιες εκφράσεις σε αυτά τα είναι α, α, ε, απλοϊκές και μη αποδεδειγμένες και χρειάζεται από το Προεδρείο κάποια ακριβή στοιχεία όσον αφορά τα σχετικά κόστη. Επίσης, με εκπλήσει ότι βλέπω στο τμήμα 6 ότι μια αλλαγή στη συνθήκη μπορεί να είναι απλή και γρήγορη διαδικασία. Η δική μου εμπειρία δεν λέει κάτι τέτοιο. Και νομίζω πως είναι σημαντικό Εμείς είμαστε ευαίσθητοι όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων καθώς και την ε, ποιότητα των ε, των ε, νόμων. Εμείς προετοιμαζόμαστε για μία μη απλοποιημένη διαδικασία για αυτό το θέμα, αλλά ένα συνολικό πακέτο προτάσεων που θα ενημερώνει την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία για την επόμενη συνέλευση που πιστεύω θα ξεκινήσει την άνοιξη του του 2015 θα είναι κάτι που θα πρέπει να το προετοιμάσουμε από τώρα. Και αυτό σημαίνει να σκεφτούμε όχι μόνο το θέμα του Στρασβούργου και του Κοινοβουλίου, αλλά και το θέμα της έδρας των άλλων θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων συμπεριλαμβανομένες μιας πιθανής αναθεώρησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που θα καθορίζει την έδρα, την, το τόπο μάλλον της κοινοβουλευτική έδρα. Επίσης, επειδή πρόκειται για ένα πακέτο ένα κατάλογο που προετοιμάζουμε θα πρέπει να ιεραρχήσουμε την ατζέντα του Κοινοβουλίου. Βέβαια, για κάποια θέματα είναι πολύ σημαντικό, αλλά για άλλα λιγότερο. Και σίγουρα είναι θέματα τα οποία θα μπουν στην έκθεση, την οποία θα εξετάσουμε την επόμενη φορά. Θα πρέπει να είναι στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρόντς, τέλος. Εγώ είμαι υπέρ τη μια έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη στιγμή που υπάρχει, μόνο και μόνο επειδή περιορίζει το κόστο. Έπειτα δεν θα σιωπήσω για το πού θα πρέπει να είναι. Πιστεύω πω θα πρέπει να είναι στι Βρυξέλλε και εν μέρη γιατί είναι πιο εύκολη στην πρόσβαση και δεύτερον γιατί το εκτελεστικό βρίσκεται εδώ για έλεγχο και για συναπόφαση από την άλλη πλευρά. Για τα διαδικαστικά ωστόσο δεν πιστεύω πως το Κοινοβούλιο εν γέννη θα πρέπει να επιτρέπεται να αποφασίζουν πού θα ε, εδρεύουν γιατί όπως είπε ο κ. Γκολτιέρη αυτό είναι θέμα συνταγματικό στη χώρα αυτή, στα κράτη δηλαδή ανήκει και κατά αναλογία πρότεινε να υπάρξει ένα θέμα τέτοιο στη συνθήκη. Η δική μου διαφωνία με τα συντάγματα της Ένωσης δεν ε, αλλάζει το θέμα ότι θα πρέπει να είναι κάτι το αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο με μια συνθήκη. Επίσης δεν είμαι ευτυχής με την ιδέα να θεωρούνται τα κοινοβούλια πλανόδια, τροχόσπιτα, τροχοβίλες που θα μπορούν να μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο ανάλογα από το, τι θα τους καπνίσει κάθε φορά. Λοιπόν, 2008 νομίζω ή 2007 ελήφθη απόφαση για μετακίνηση προσωρινά στο Βρυξέλλες, στις Βρυξέλλες λόγω δομικών προβλημάτων που υπήρχαν στο Στρασβούργο και εκεί δημιουργήθηκε ένα κάποιο προηγούμενο. Ε, Χθε δεν έλαβα απάντηση στην ερώτησή μου, αλλά αυτό που ήθελα να γνωρίζω είναι ποια ήταν η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για να νομιμοποιηθεί η απόφαση του 2007 και 2008 ή ο μηχανισμός, ποια, τι βρήκατε για να το νομιμοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, ο Γκέραλτ Χέφνερ. Να παρέμβει όπως ζήτησε από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ γόνιμη η συζήτηση και κατά τα άλλα η ακρόαση επίσης εξαιρετική και πολύ διαφοροποιημένη και στις τοποθετήσεις των εισηγητών αλλά και στη συζήτηση ε, με τους εμπειρογνώμονες. Σπάνια έχω δει τέτοια ε, συζήτηση σε ακρόαση που μέσα σε δύο ώρες ακούσαμε δύο εμπειρογνώμων, τέσσερις εμπειρογνώμων, 13 μέλη της Επιτροπής. Είχαμε πολύ λίγο χρόνο να την προετοιμάσουμε, αλλά την προετοιμάσαμε σε μεγάλο βάθος και πολύ μεθοδικά. Και οι εμπειρογνώμες ξαναπήραν το λόγο μετά για να κλείσουν. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα ήθελα να ε, πω ε, τα εξή σε δύο μιλητέ. Στην κυρία Λεξίμερα αναλώσατε πάρα πολύ χρόνο να επικρίνετε την πρόσκληση. Το κάνατε και σε μένα προσωπικά. Εγώ μπορώ να επαναλάβω ό,τι σας είπα, δεν θα το κάνω, θα χάσουμε χρόνο. Αν αυτό είναι το πρόβλημα και θέλουμε να τσακωθούμε γι' αυτό, πραγματικά με εκπλήσει. Εμένα θα με ενδιαφέρει πιο πολύ το θέμα της έδρας και η ουσία, γιατί προσπαθούμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να αφήσουμε τελείως ε, ανοιχτό το ενδεχόμενο της τελικής απόφασης για μία έδρα. Φαίνεται δεν σας έχω πείσει σας, έχω πείσει όλους τους άλλους. Ελπίζω να μπορέσω να σας κερδίσω και σας. Ε, το θέμα δεν είναι η Βρυξέλλη Στρασβούργο, αλλά να έχει τη δυνατότητα το Κοινοβούλιο να το αποφασίζει είτε μόνο του, είτε εν πάση περιπτώσει να συναποφασίζει. Για μένα ακούσαμε σχετικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από τον κύριο Γκουαλτιέρη και από τον κύριο Βίλαντ ε, και από τον κύριο Νταφ. Τελικά με το έγγραφο εργασίας απλώς υπονοούμε τη διαδικασία, δεν το έχουμε συγκεκριμενοποιήσει ούτε ξεκαθαρίσει όσο θέλουμε να το κάνουμε στην έκθεση. Και για το σημείο 7, την κριτική σας, με την ίδια διαδικασία, το same procedure είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο να παρερμηνευτεί δεν θέλουμε μια απλουστευμένη διαδικασία, ούτε ταχεία, αλλά η μόνη δυνατή διαδικασία είναι αυτή που λέγουμε, να είναι ένα τμήμα μιας μεγαλύτερης αλλαγής της συνθήκης που θα χρειαστεί οπωσδήποτε συντακτική συνέλευση και στη συνέχεια διακυβερνητική διάσκεψη. Άρα το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή μια δέσμη ετοιμάζει, ένα πακέτο με διάφορα θέματα. Αυτό το είπαμε και για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θέματα που απασχολούν το Κοινοβούλιο και που θα θέσει σε μια συντακτική συνέλευση που οπωσδήποτε θα χρειαστούμε μετά τις επόμενες ευρωεκλογές. Και ορισμένοι λέγουν ότι η έδρα θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο των εδρών των άλλων θεσμικών οργάνων. Θα ήμασταν αφελείς αν το παραγνωρίζαμε κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ σφάλμα τώρα στο ένα έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βάλουμε κάτι το οποίο αργότερα θα είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Τα συγκεκριμένα να τα περιορίσουμε μόνο στα δικαιώματα ε, του Κοινοβουλίου και την αυτοοργάνωση. Να μην βάλουμε στη δική μας έκθεση τώρα ζητήματα εδρών άλλων θεσμικών οργάνων. Αυτά. Επί της ουσίας, ε, να πούμε για τα νομικά, για τα πολιτικά. Κάποια στοιχεία αριθμητικά αναφέρθηκαν. Και πάλι, κυρία με μένα τι με ενδιαφέρει, δεν θέλω να διαπληκτιστώ μαζί σα για τα αριθμητικά στοιχεία. Εβδομάδε ολόκληρε προσπαθήσαμε να βρούμε αριθμητικά στοιχεία ξεκάθαρα και με εκπλήσει που το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει υπολογίσει το κόστο, Νομίζω ότι είναι εύκολο σχετικά. Ε, οι ε, βουλευτές υποβάλλουν δικαιολογητικά και γνωρίζουμε ποιο είναι το κόστος ταξιδίων. Τώρα έχουμε βάλει αυτά τα στοιχεία, κάποιοι τα αμφισβητούν, τα αντικρούν, αυτά ακούμε. Λοιπόν, είναι έγγραφο εργασίας, επαναλαμβάνω. Ένα έγγραφο εργασίας παραθέτει και απαριθμεί ε, τα επιχειρήματα. Στην έκθεση δεν θα διαπλεκτιστούμε για αριθμούς, ούτε θα αποφασίσουμε, αλλά θα ψάξουμε ε, τη νομική οδό όσο και την πολιτική αξιολόγηση. Οπότε ας μην ε, ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το θέμα. Επίσης με εξέπληξαν διάφορα άλλα πράγματα. Μας προσάπτεται ας πούμε κυρία Λεκρύπ ότι θέλουμε να κάνουμε διακρίσεις. Ότι ε, το έγγραφο αυτό είναι ε, αμφισβητήσιμο και αμφισβητούμενο ότι συζητάμε για το χρώμα των ταξί και δεν είναι το επίπεδο αυτό της Επιτροπής μας. Πού τα λέει αυτά το έγγραφο εργασίας. Ας μην ρίξουμε τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο τις άλλες τοποθετήσει ευχαριστώ πολύ. Τελικά, τι θα κληθούμε να αποφασίσουμε, το είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι. Για μένα παραμένει ακόμα ανοιχτό. Στο τέλος, το κοινοβούλιο μόνο του θα θέλουμε να ζητάμε να παίρνει αυτή την απόφαση ή το κοινοβούλιο στα πλαίσια μια συντεταγμένης διαδικασία σε συναπόφαση με το Συμβούλιο. Και έχει νόημα να πει το Κοινοβούλιο ότι εμείς θέλουμε να είμαστε σε θέση να συναποφασίζουμε, να συνδιαμορφώνουμε την απόφαση αυτή. Το δρόμο δεν τον έχουμε βρει, θα πρέπει να το διαπραγματευτούμε και σε μεγάλο βάθος εδώ στην Επιτροπή μας. Τελευταίο. Θα ήθελα να διατηρήσω αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, παρακαλώ, να με το νομικό θέμα, με το συνταγματικό, το θεσμικό και όχι αποφαινόμαστε υπέρ της μιας ή της άλλης έδρας. Παρακαλώ να κρατηθεί εκεί η συζήτηση αυτή και χαίρομαι που έγινε. Είναι θέμα δημοκρατικό, είναι ένα θέμα συνταγματικό, συνθήκων, δεν είναι υπέρ κατά μιας χώρας, μιας πόλης ή ό,τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much uh, for your... Uh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας ε, είπατε. Ε, Πράγματι λοιπόν εχθές είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και εχθές ζήτησα από τη γραμματεία να με ε, να πάρει τα έγγραφα και τις ομιλίες ε, των συναδέλφων σε γραπτή μορφή, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα είναι χρήσιμο για τους δύο αλλά και για όλους μας που παρακολουθήσαμε το θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Κλείνει αυτό το θέμα. Επανήλθε εδώ και ο κύριος ε, Κασίνη και θα συνεχίσει εκείνος ε, να προεδρεύει για την επόμενη έκθεση εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Bene, πολύ ωραία. Ξεκινάμε ε, επαναλαμβάνω, ξανααναλαμβάνω μάλλον την Προεδρία. Η κυρία Γκουτσέκ τα έκανε πάρα πολύ καλά. Μάι, με συγχωρείτε. Έχουμε λοιπόν το χρόνο ε, αρκετό για να περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχει σχέση με την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Κατ' ουσίαν ε, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ενημερωθούμε για το τι ακριβώς ελέγχθη στον τριμερή διάλογο. Σύμφωνα με το άρθρο 70, κυρίως μετά την έκθεση Γκορέρο, προβλέπεται η διαπραγματευτική ομάδα να αναφέρεται μετά από κάθε συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου στην αρμόδια επιτροπή. Θα θυμάστε λοιπόν ότι η έκθεση της κυρίας Γιαννάκου εγκρίθηκε στις 15 Απριλίου. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έλαβε χώρα στις 16 Απριλίου στο Στρασβούργο και μία δεύτερη συνεδρίαση στις 15 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Το βασικό λοιπόν θέμα που συζητήθηκε ήταν τελικά ποιο, όργανο είναι αρμόδιο για να καταγράψει τα πολιτικά κόμματα. Σε εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσαμε ότι το Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο για την καταχώρηση των πολιτικών κομμάτων και την ε, αναγνώρισή τους. Την εγγραφή τους και την αναγνώρισή τους. Αυτό λοιπόν το στήριξε η Επιτροπή και θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα αυτοματισμού στην ε, εγγραφή. Θα ήταν άσχημο ένα όργανο όπως ε, τον ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην είναι ένα όργανο το οποίο να μπορεί να κρίνει για τις ε, απόψεις που δημορφώνται σχετικά με τα κόμματα και σε σχέση με την ελευθερία, την ενημέρωση, ε, να μπορεί δηλαδή να αποφασίσει σε επίπεδο αρχής σχετικά με τα κόμματα. Από τις, ε, ή μάλλον στη διάρκεια των συζητήσεων καταβλήθηκαν προσπάθειες να διατηρηθούν οι αρμοδιότητες σχετικά με την εγγραφή στο Κοινοβούλιο. Εκείνο όμως το οποίο προέκυψε ήταν ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις πολιτικοποιούνται στο μέγιστο βαθμό και κατόπιν τούτου ε, θα πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή σοφών ή κάποιος άλλος ο οποίος να μπορεί να αποφαίνεται ως προς την ε, τήρηση των αρχών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με ένα πολιτικό σχηματισμό. Νομίζω όμως ότι η συγκήτριά μας η κυρία Γιαννάκου μπορεί να μας δώσει περισσότερες ε, πληροφορίες από αυτού του θέματος. Παρακαλώ κύριε Γιαννάκου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι έγινε, <coughs> έγιναν συναντήσεις που είπατε καθώς και ένας τεχνικός διάλογος μεταξύ της Γραμματείας και των υπηρεσιών των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με το Συμβούλιο φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση παρά το γεγονός ότι ορισμένες χώρες ακόμα δεν έχουν πάρει σαφή θέση σε ορισμένα ζητήματα υπάρχει διάθεση από την Ιρλανδική Προεδρία να τελειώσει εντός της Ιρλανδικής Προεδρίας η υπόθεση αυτή. Απ' την άλλη πλευρά ε, θα πρέπει να ε, σημειώσω ότι όλοι τονίσαμε ότι πρέπει να κατασυγαστούν οι φόβοι του Συμβουλίου και ότι και εμείς στο Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι η εγγραφή των είναι αυτόματη και πρέπει να είναι ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές. Προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να κατασυγαστούν οι ανησυχίες του Συμβουλίου. Την επομένη εβδομάδα θα επαναληφθεί εξ όσων γνωρίζω μία συνάντηση τεχνικού χαρακτήρα ε, χωρίς την παρουσία των βουλευτών αλλά και εγώ την επόμενη εβδομάδα θα ζητήσω να βρεθούμε μαζί οι συντονιστές οι Σάντο συγγνώμη, και οι συντονιστές για να κάνουμε μια, να ξαναβούμε λίγο από την αρχή την όλη υπόθεση. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ελπίδες όπως είπε και ο Πρόεδρος. Ο Τρίλογος θα επαναληφθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Στρασβούργου. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι το περίφημο θέμα για, την, ε, ε, για το σεβασμό των βασικών αρχών και αξιών της Ένωσης μπορεί κάλλιστα και αυτό να τοποθετηθεί με τελείως ε, ε, τυπικό τρόπο μέσα από μια application form ε, η οποία θα δίδεται από την υπηρεσία αυτή την όποια υπηρεσία που και εμείς θέλουμε να εγκατασταθεί στο Κοινοβούλιο ώστε να μην δημιουργείται πάλι ζήτημα κάποιου πολιτικού κριτηρίου ή κάποιας πολιτικής εμπλοκής. Φυσικά επαναλάβαμε τη θέση μας ότι δεν θέλουμε περισσότερα χρήματα για τα κόμματα σε καμία περίπτωση, άρα δεν θέλουμε να ξοδέψουμε και χρήματα για δημιουργία νέων οργάνων και οργανισμών. Γιατί είχε υπάρξει από την αρχή στο Συμβούλιο κάποια ιδέα για ένα νέο agency. Έχουμε τονίσει ότι επιζητούμε ένα τρόπο να είναι ανεξάρτητα και διοικητικού χαρακτήρα τα όργανα για αυτόματη εγγραφή των κομμάτων αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε νέους οργανισμούς, νέα έξοδα και νέα συστήματα να δημιουργήσουμε. Έτσι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε όπως είπα μια τεχνική συνάντηση, μια συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές ε, για να συνεννοηθούμε για το ε, τι έχει γίνει μέχρι τώρα και στο Στρασβούργο θα επαναληφθεί ο τρίλογος επίσημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκουρμάη ζήτησε το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως ε, Ξέραμε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα ήταν εύκολες και οι πρώτες συνεδριάσεις το επιβεβαίωσαν. Παρ' όλα αυτά σημειώσαμε κάποια πρόοδο και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέδειξε τη βούλησή του να μετακινηθεί από την αρχική του θέση και να βρει, να αναζητήσει ένα συμβασμό ικανοποιητικό για όλους. Και νομίζω η συγγήτρια εργάστηκε πολύ σκληρά. Ε, προσβλέπω σε μια παρεμφερή κίνηση από το Συμβούλιο και ελπίζω στην άλφη του Συμβουλίου που παρήσατε εδώ να έλαβαν το μήνυμα. Όσον αφορά το θετικό ε, μήνυμα τη χθεσινή συνεδρία, είναι ότι επιτέλου υπάρχουν συγκεκριμένε ε, προτάσει μέσα από τα αποκαλούμενα non-paper. Πρέπει λοιπόν ταχύτατα να ξανασυναντηθούμε για να ε, στείλουμε και εμεί το δικό μα το μήνυμα, Κυρίω επειδή όπω είπε και η Μαριέτα, οι Ιρλανδοί θέλουν και άλλη συνεδρίαση υπό την Προεδρία του, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στην επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Όσον αφορά τώρα στι προτάσει που έχουν κατατεθεί, εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή ε, με βάση, μάλλον στην τελευταία συναντρίαση και μετά από την πρόταση του κ. Κωσίνη, η Επιτροπή ε, θεωρεί ότι αυτά που προτείνει το Συμβούλιο είναι πολύ καλύτερα. Δηλαδή ένα είδος ε, διαδικασίας συναπόφασης, αλλά στην περίπτωση της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ αυτό που προτείνεται κατά την άποψή μου είναι πολύ προτιμότερο, δηλαδή να περνάει το θέμα μέσα από την Επιτροπή των Σοφών και όχι να υπάρχει κάποιος αυτοματισμός. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην προκύψει μια επίπονη διαδικασία, κυρίως ε, δεν είναι και σαφής η τελική υπεραξία που θα προκύψει. Βλέπω ότι το έγγραφο της Κομισιόν περιλαμβάνει αρκετές ρήτρες ασφαλείας για να μπορεί το Κοινοβούλιο να ασκήσει τα δικαιώματά του. Αν λοιπόν θέλουμε να αποφύγουμε σύγκρουση συμφερόντων, πάντων δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια δημοκρατική νομιμότητα που δεν έχει κανένας άλλος ευρωπαϊκός θεσμός και το είπε αυτό και η Μαριέτα. Αυτών όλων λεχθέντων ελπίζω ότι το Συμβούλιο τελικά θα προτείνει μια συμβαστική πρόταση και θα μπορέσουμε να περάσουμε στις επόμενες φάσεις της συζήτησης. Λυπάμαι όμως που εξακολουθούμε ε, να μην έχουμε άλλες απόψεις από άλλα κρατημέλη. Κατανοούμε βέβαια ότι φοβούνται τις επιπλέον επιπτώσει αυτού του κανονισμού στην ε, δική του την εθνική νομοθεσία και διαφωνούν με την ε, συμμετοχή πολιτικών κομμάτων σε εθνικά ε, δημοψηφίσματα ακόμα και για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανησυχίες πρέπει να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία αγαπητή εισηγήτρια κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστούμε την κυρία Γκουρμά. Ο κύριος Νταφ έχει το λόγο. Πρόεδρε, νομίζω ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, κινούνται κάπως τα πράγματα, ιδιαίτερα από πλευράς Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται πρόθυμη να προχωρήσει, να βοηθήσει και περιμένουμε μια σαφή εξήγηση ακόμα για το νομικό καθεστώς ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. στο δίκαιο της Ένωσης. Και πώς θα μπορεί να λειτουργεί ένα πολιτικό κόμμα εντός μιας προεκλογικής εκστατείας για τις προεκλογές. Σε κάποιο κράτος μέλος. Δηλαδή, ποια είναι τα πλεονεκτήματα που θα έχει ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Εάν υποκαταστήσουν το καθεστώς, ας πούμε, του Εθνικού Κόμματος υπό Βελγικό Δίκαιο. ως προς το νομικό καθεστώς, το ευρωπαϊκό, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν κάποιες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, αλλά ακόμα δεν τις έχουμε λάβει από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι για να προχωρήσουμε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο την ακριβή φύση την ακριβή φύση όμως αυτής της Επιτροπής Σοφών και το μέγεθος και τη σύνθεσή της ε, και την εντολή της και τις εξουσίες της και τον τρόπο και τη μέθοδο εργασίας της. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή στους τριμερείς διαλόγους που είχα ε, συμμετάσχει γίνεται μια γενική και αόριστη συζήτηση ε, χωρίς κοινή συνισταμένη. Ε, και δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει ούτε προχωρεί έτσι η συζήτηση, ούτε τελικά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη πολιτική συνένεση σε αυτό το θέμα που είναι τόσο λεπτό και ευαίσθητο. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν το Συμβούλιο ως συνομοθέτης θα είναι τμήμα της απόφασης η απαγόρευση ενός πολιτικού κόμματος. Η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου φαίνεται να φρονεί ότι κανονικά θα πρέπει να συμμετέχει το Συμβούλιο σε μια τέτοια απόφαση, διότι ο γενικός κορμός, ας πούμε, της συνταγματικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υπάρχει ε, ε, μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των ε, νομοθετών. Και, ε, θα ήθελα να ακούσω, βέβαια μου φαίνεται λογική αυτή η πρόταση, αλλά θα ήθελα να ακούσω τις αντιδράσεις ε, για αυτό το θέμα. και ε, το εισηγητή σε ό,τι αφορά τα δημοψηφίσματα. Τι ρόλο θα παίζουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σε εθνικά δημοψηφίσματα για ευρωπαϊκά θέματα. Και εγώ πιστεύω ότι συμφωνούμε εδώ ότι και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε ε, στην αντιπροσωπεία μας, στον τριμερή διάλογο, μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να τραβήξουμε αυτή τη θέση. Αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και αίτημα. Grazie, onorevole Um, Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος είπε ότι ε, πρέπει να αποπολιτικοποιήσουμε το όλο θέμα της ε, εγγραφής και αναγνώρισης ε, των κομμάτων. Εάν όμως το όλο θέμα έχει συνταχθεί από πολιτικούς, η απόφαση σχετικά με την εγγραφή και την αναγνώριση γίνεται πλέον μια αντικειμενική απόφαση με βάση όμως υποκειμενικά κριτήρια. Δηλαδή τα περισσότερα ολοκληρωτικά συστήματα ε, φέρνουν σε μειονεκτική θέση τους αντιπάλους μέσα από τους δικούς τους τους κανόνες. Επιπλέον σήμερα το πρωί ο πρόεδρος κάνοντας ε, την παρουσίαση από τις συνεδρίες των συντονιστών και ελπίζω να κατάλαβα καλά μας είπε ότι υπάρχουν ήδη δύο συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη διαγραφή ενός ε, κόμματος από το Μητρό που δεν μπορεί όμως να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή γιατί δεν υπήρχαν και οι όροι για να εγγραφεί. Αν αυτό ισχύει, τότε αυτό δεν είναι καλός ιονός για τις ε, μελλοντικές αποφάσεις από πολιτικοποίησης, γιατί ε, μπορεί και κάποιοι να κάνουν ε, αιτήσει χωρίς να αναφέρουν κανένα άλλο λόγο. Ελπίζω να κατάλαβα καλά. Ο κύριος ε, Χέφνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα είμαι σύντομος ε, και θέλω να πω κάτι το οποίο έχει σχέση με αυτά τα οποία ήδη αναφέρθηκαν. Διότι κατά τα άλλα, όσον αφορά τη διαπραγματευτική ομάδα, έχουμε ξεκινήσει τη συζήτησή μας και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έχουμε φτάσει σε τέτοια φάση έτσι ώστε από το Συμβούλιο να προβάλλονται, να διατυπώνονται συγκεκριμένε προτάσει. Κατανοώ βέβαια ότι το Συμβούλιο χρειάζεται κάποιο χρόνο, αλλά ελπίζω πλέον να προχωρήσει με ταχύ ρυθμό. Κοιτάξτε, για μένα όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λόγω των υφιστάμενων κανονισμών αντιμετωπίζουμε δυσκολίες οι οποίες κατέστησαν σαφείς με τα λίγα που είπε στην αρχή ο πρόεδρος, όταν ξεκίνησε δηλαδή η συνεδρίασή μας. Δεν θέλω να πω τίποτα περιττέρω για το ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο και ποιες είναι οι δυσκολίες. Μόνο που θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο η εμπειρία που συγκεντρώνουμε να συμπεριληφθεί ε, σε αυτά που θα συζητήσουμε στο μέλλον. Και αν φανεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία, μια διαδικασία η οποία θα είναι όσο πιο μακριά γίνεται από πολιτικές ε, επιρροές και αποφάσεις, μια απόφαση που θα βασίζεται σε γεγονότα και νομικά ε, θα είναι αδιαμφισβήτητη. Αν τα επιθυμούμε όλα αυτά, νομίζω ότι μέχρι τώρα ε, δεν έχουμε μεριμνήσει προς αυτήν την κατεύθυνση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε μια τέτοια διαδικασία. Και επίσης όσον αφορά ε, το ποιος ε, στο Κοινοβούλιο θα ασχολείται με ποιο τρόπο για αυτά τα θέματα. Και όσον αφορά στο ρόλο ε, την σύνθεση και την κατανόηση των περίφημων σοφών, των eminent persons, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξανακάνουμε μία συζήτηση έτσι ώστε αυτοί που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στον τριμερή διάλογο να ενημερωθούν πλήρως για αυτά τα οποία αποφάσισαν οι συντονιστές στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις των συντονιστών. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλος ε, το λόγο. Θέλω να σας πω ότι εγώ στον τριμερή διάλογο στο τέλος της ε, συνάντησης, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπάθησα να παροτρύνω σε ταχύτερο ρυθμό στις ε, συζητήσεις. Συμφώνησα βέβαια με την άποψη της εισηγητριάς μας, της κυρίας Γιαννάκου, να κατατεθεί μία έκθεση στην Επιτροπή. Προσπάθησα δηλαδή να εξηγήσω καλύτερα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινώντας από την αρχή, από την αρχή της ε, αρχής ε, ε, του συνέρχεστε. Ένα πολιτικό κόμμα είναι νομοθετικής φύσεως θέμα, άρα δηλαδή απαιτεί και την ισχυρή συνύπαρξη των δύο νομοθετών. Αυτό βέβαια είναι κάτι αυτονόητο. Εμείς προσπαθούμε να ορίσουμε ένα ημιαυτόματο θέμα όπου όχι ένας ε, θεσμός αλλά μια συγκεκριμένα υπηρεσία του Κοινοβουλίου, όχι ένας οργανισμός αλλά μια υπηρεσία του Κοινοβουλίου θα ρυθμίζει αυτά τα θέματα ε, ε, τι επιτρέπεται με βάση το καταστατικό, το ποια θα πρέπει να είναι η έδρα. Αυτά δηλαδή τα τυπική σε φύσεως θέματα ε, μπορούν να γίνουν, να διευκρινιστούν πάρα πολύ εύκολα. Όσον αφορά τώρα την ταύτιση με τις αξίες, αυτό σαφώς και είναι ένα πολιτικής φύσεως θέμα, εκεί πολιτικοποιείται το θέμα. Άρα δηλαδή θα υπάρχει μια επιτροπή σοφών που θα αποφασίζει κατά πόσον πρέπει ένα κόμμα να εγγραφεί και να αναγνωριστεί. Εάν δηλαδή υπάρχει κάποιος που θα μπορούσαν να είναι μια ομάδα βουλευτών που θα θίξουν το θέμα. Εγώ πιστεύω, όπως σας είπα, ότι θα υπάρχει αυτή η Επιτροπή των Σοφών που θα μπορούν να τοποθετηθούν σχετικά με ερωτήματα που θα τεθούν. Είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Νταφ, σε σχέση με την Επιτροπή ότι το κατσατικό αναφέρει ή ότι θα πρέπει να, να σεβόμαστε τις αρχές του κατσατικού για να διεκδικήσουμε την εγγραφή και την καταχώρηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα αποφαίνεται η Επιτροπή των Σοφών. Η κυρία Γιαννάκου ε, πολύ σωστά λέει ότι η άποψη των σοφών θα είναι συμβουλευτική και δεν θα είναι εκείνη που θα καθορίζει απολύτως τα θέματα. Αυτά λοιπόν έχουν τεθεί επιτάπητος. Δεν ξέρω τελικά αν θα κατορθώσουμε να εμφανιστούμε με μία φωνή και αν θα έχουμε και την στήριξη της Επιτροπής. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε και το Συμβούλιο επί του θέματος. Ελπίζω να ερμήνευσα σωστά την άποψη, την κυρίαρχη άποψη της Επιτροπής και έτσι θα προχωρήσουμε στο μέλλον στον τριμερή διάλογο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος της ε, Στοκχόλμης. Τώρα απευθύνομαι στο Συμβούλιο. πριν τεθεί ε, το πρόγραμμα η συνθήκη σε εφαρμογή, η δική μας επιτροπή ενέκρινε μία έκθεση η οποία αφορά ακριβώς στην ε, εφαρμογή του προγράμματος της ε, Στοχόλμης. Για πρώτη λοιπόν φορά εφαρμόζεται το άρθρο 51 τη συνεργασία ανάμεσα στις ε, επιτροπές, ε, την Νομική Επιτροπή, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Να γίνει λοιπόν μια ενδιάμεση έκθεση, ένας έλεγχος του τι έχει λάβει η χώρα, έτσι ώστε να δώσουμε κάποιες ενδείξεις ε, για μελλοντικές νομοθετικές πράξεις, αλλά και για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε να κάνουμε λοιπόν αυτή την αξιολόγηση και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα αίτια. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο προτείναμε μία ερώτηση προς την Επιτροπή και προς το Συμβούλιο για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Και μας είπαν ότι έχουν γίνει πάρα πολλά, ακόμα βέβαια ε, διάφορα υπολείπονται. Μας απαρίθμησαν ε, τους κανονισμούς, τις προτάσεις που έχουν εγκριθεί, αλλά υπάρχει και ένας κατάλογος πραγμάτων που δεν έχουν γίνει. Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Το δικό μου το πρόβλημα, και εδώ ζητώ τη συμβουλή σας, είναι το εξής. Εγώ έχω στα χέρια μου έγγραφα εργασίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Πρόκειται λοιπόν για έγγραφα τα οποία απαριθμούν το τι έχει γίνει και το τι πρέπει να γίνει. Και μάλιστα με κάποιο κριτικό πνεύμα επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι δεν έχει προχωρήσει ορισμένα θέματα, αλλά και το Κοινοβούλιο, γιατί δεν έχει εφαρμόσει τις προτάσεις της Επιτροπής σε ορισμένα θέματα. Ε, υπάρχει ο κατάλογος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης αφορά το χώρο ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας που περνάει από το τρίτο πυλώνα στην διαδικασία και αρμοδιότητα νομοθεσία. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που πρέπει να εξετάσουμε. Έχουμε λοιπόν δύο έγγραφα εργασίας που όπως σας είπα απαριθμούν το τι έχει γίνει και το τι ακόμα υπολείπεται. Εδώ το πρόβλημά μου είναι και θέλω να με συμβουλεύσετε είναι κατά πόσον και η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να προετοιμάσει το δικό της το έγγραφο εργασίας. Όμως νομίζω ότι δεν ενδείκνεται και πολύ κάτι τέτοιο γιατί αν θέλουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που μας έχει τεθεί ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε ήδη κατά την επόμενη Επιτροπή Άρα το να, καταστήσουμε, να καταρτήσουμε ένα έγγραφο εργασία δεν ξέρω μήπως θα καθυστερήσουμε. Ίσως καλύτερα να συνεργαστούμε με τους δύο άλλους συγητές που έχουν ήδη συντάξει ένα έγγραφο και αυτό το τελικό έγγραφο να το υποβάλουμε σε συνεδρίαση των τριών επιτροπών. Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου νομίζω ότι είναι καλύτερο να διαλέξουμε αυτό το δεύτερο δρόμο. Βέβαια θα ήθελα να κατανοήσω καλύτερα τελικά τι πρέπει να κάνω εγώ σε σχέση με την σύνταξη της έκτασης ε, και το πώς πρέπει να συνεργαστούμε με τους άλλους δύο εισηγητές. Δεν είναι Μάλλον, να το πω αλλιώ. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων λένε ότι στον εμπορικό τομέα έχουμε κάνει αυτό ή στον άλλο τομέα πρέπει να κάνουμε το Β ή στον τομέα των θεωρήσεων έχουμε κάνει τα εξή ε, στην ε, υπεράσπιση των συνόρων. Έχουμε τη Frontex αλλά δεν αρκεί αυτό. Έχουμε το Schengen αλλά δεν διευρύνθηκε αρκετά. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη σειρά θεμάτων που αναφέρεται. Εγώ όμως νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι αφορά ιδιαίτερα τη δική μας την Επιτροπή. Η δική μας Επιτροπή έχει συγκεκριμένα επιχειρήματα τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της Εκόλμης. Παραδείγματο χάρη, η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την διαφύλαξη των θεμελιωδών ελευθεριών. Εκεί βρισκόμαστε στο τελικό φάση, στην τελική φάση σύνταξης ή ε, για την πρωτοβουλία των πολιτών. Και αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο επιχείρημα της δικής μας Επιτροπής. Ίσως μπορούμε επίσης να αναφερθούμε και στις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα τη δική μας Επιτροπή. Σήμερα μάλιστα συζητήσαμε για τις απόψεις ε, που τρέχουν τώρα ε, σχετικά με την ε, διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα και με τις ε, σχέσεις του Κοινοβουλίου με τις ε, επιτροπές ε, και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όλα αυτά τρέχουν. Να δούμε λοιπόν το τι πρέπει να πει ο εισηγητής ο δικός μας στη συνεργασία με τους δύο άλλους εισηγητές. Εμείς ασχολούμεθα με το συνολικό, το σφαιρικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κατά νου το τι έχει γίνει και το τι υπολείπεται ακόμα στα διάφορα σημεία του προγράμματος της Στοχόλμης. Θεωρώ λοιπόν ότι κάτω από αυτό το πρίσμα αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να δώσουμε σημασία στην αρμοδιότητα της συναπόφασης, συνομοθεσίας. Αυτό είναι κάτι πολύ καινούριο. Προέκυψε από τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας και αυτό το θέμα αφορά όλα τα επιχειρήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης. Ε, υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις σχετικά με τις ε, διαπραγματεύσεις για την πρώτη ανάγνωση, κατά πόσον πρέπει να επιταχύνονται οι διαδικασίες. Για όλα αυτά θα ήθελα να ακούσω τη δική σας την άποψη. Έχει λοιπόν ζητήσει το λόγο Συνάδελφο Στέιν, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι εδώ σκιώδης στη συγκήτρια των φιλελευθέρων. Και σε σχέση με τη διαδικασία θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνούμε με τη δεύτερη λύση που προτείνατε. Το βρίσκω λίγο κρίμα όμως που είμαστε πάλι υπό τέτοια χρονική πίεση. Διότι είναι γεγονός ε, ότι ε, ε, ε, γίνεται λόγος για ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά ποια ενδιάμεση, είναι σχεδόν οριστική αναθεώρηση, τελική αυτή. Ε, για τον απολογισμό λοιπόν θα χρειαζόμασταν λίγο περισσότερο χρόνο. Αν σκεφτεί κανείς ότι αγγίζουμε περίπου το τέλος της θητείας μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια τελική αξιολόγηση έτσι οριστική, διότι έτσι περί το τέλος δεν νομίζω να αποφασιστούν και πάρα πολλά καινούρια. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το πρόγραμμα της Στοχόλμης, το είχαμε περάσει υπό τεράστια πίεση. Νομίζω ο Ούγγρος συνάδελφος πήρε το κείμενο στα Ουγγρικά κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, για να καταλάβετε. Και γι' αυτό έχει σημασία, πιστεύω, για τους πολίτες όταν έχουμε ένα τέτοιο σημαντικό πρόγραμμα και τόσο φιλόδοξο να μην το περνάμε άρον-άρον για να δούμε τώρα τι έχει ε, εφαρμοστεί και όχι μόνο επιμέρους σημεία, αλλά να κάνουμε και μια στατιστική καταγραφή πώς από όλα αυτά τα σημεία που περάσαμε τόσο βιαστικά εφαρμόστηκαν, με ποια ε, ποιότητα, πόσο καλά εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, όχι μόνο αριθμητικά τα μισά, αλλά ουσιαστικά, ποιοτικά, τι έχουμε εφαρμόσει από αυτά που αποφασίσαμε. Εδώ συνεργασία μεταξύ των τριών επιτροπών ήταν και πιστεύω ότι και η δική μας επιτροπή ε, σωστό είναι να συμμετέχει και να το ε, κοιτάξει και να το μελετήσει ουσιαστικά και όχι έτσι εμπαρόδο. Ήταν ένα πρόγραμμα πολιτικό και χρειάζεται και ένας πολιτικός απολογισμός. Αυτό το οφείλουμε στους πολίτες ε, που θέλουν να δουν τι πολιτικούς στόχους θέσαμε και τι υλοποιήσαμε. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω εικόνα. Ε, ήταν 150 σημεία, πάρα πολλά. Δεν μπορώ. Ε, πρέπει να, τελικά να καταλάβουμε τι επιτύχαμε και τι δεν επιτύχαμε. Um, ναι, και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί πρέπει να γίνουν όλα αυτά τόσο βιαστικά. Εάν θέλουμε σοβαρά να δουλέψουμε, πρέπει να τα δουλέψουμε και σωστά. Από την προοπτική της ΑΦΚΟ, Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσουμε αν οι εξαιρέσεις των οποίων χαίρει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Ιρλανδίας κατά κάποιο τρόπο, αν έχουν περιπλέξει την νομοθετική διαδικασία και την ποιότητα του αποτελέσματος. του ευρωπαϊκού δικαίου, ιδιαίτερα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την προθεσμία όπου το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προβεί σε ένα μαζικό opt-out για όλες τις νομοθεσίες πρόλης αγώνας. Νομίζω πως το συνταγματικό τμήμα αυτή τη υπόθεση, το οποίο θα, εξετάσει, θα πρέπει να εξετάσει μάλλον η ΑΦΚΟ. Και μετά, αν είναι απαραίτητο, να καταλήξει σε συμπεράσματα από το καθεστώς, την ισχύ μάλλον του καθεστώτος της σύνδεξης της μέχρι στιγμής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στον προβληματισμό μας για το τι μπορεί να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μέσω της αναθεώρησης της συνθήκης. Με άλλα λόγια, να είμαστε συνεπείς με τα όσα κάνουμε με τις άλλες εκθέσεις ε, στο τέλος της θητείας και να προετοιμάσουμε ένα τμήμα ενός καταλόγου για την επόμενη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στην συνέλευση. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να αναζητά το λόγο. Και έχουμε και ακόμα κάποια θεματάκια. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε με αυτή την παρατήρηση τη δική μου. Καταρχήν, το αίτημα για μια έκθεση τέτοιου τύπου προκύπτει από την πρωτοβουλία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, η οποία εξ αρχής πολύ βιαστικά θέλησε να κλείσει το θέμα από την αρχή. Εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και για να προβλε... προτρέξουμε αυτής της έκθεσης με μια πρώτη συζήτηση μέσω της παρουσίασης ενός αιτήματος σε μια προφορική ερώτηση που ήδη έγινε. Τουλάχιστον αρχίσαμε κάπως να το σκεφτόμαστε. Βρίσκω πως ε, και τα πράγματα τα οποία είπατε τώρα παρεμβαίνοντας είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα τα λάβω με υπόψη. Ιδιαίτερα όπως είπατε κύριε Ντάφα, είναι πολύ σημαντικές οι λεπτομέρειες. Τώρα το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Πετύχαμε μια παράταση για σε σχέση με αυτό που είχε προτείνει ε, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Δηλαδή θα πρέπει να υποβάλουμε ε, την έκθεση στην ε, εβδομάδα 3 με 10 Ιουλίου για να μπορέσουν να υποβληθούν τροπολογίες εντός του Σεπτεμβρίου, τις 3 Σεπτεμβρίου, να φτάσουμε στην αξιολόγηση των τροπολογιών στα τέλη του μήνα του Σεπτεμβρίου και να φτάσουμε στη τελική ψηφοφορία στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο. Πάνω κάτω αυτό συμφωνήθηκε με τις άλλες επιτροπές. Νομίζω πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάντως εγώ έχω υπόψη μου τα όσα είπατε, τους προβληματισμούς σας και θα προσπαθήσω προφορικά στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής να διευκρινίσω καλύτερα τη δική μας θέση στην έκθεση που θα παρουσιαστεί τον Ιούλιο έτσι ώστε και για τις τροπολογίες να μπορέσουμε να σκεφτούμε τι θα πούμε. Ευχαριστώ και περνάμε στο τελευταίο προσυζήτηση σημείο που αφορά μισό λεπτό. Ε, αφορά λοιπόν την διαδικασία έγκρισης και τους κανόνες που ισχύουν για την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σακόφσκι. Αφού συζητήσαμε το θέμα των εδρών των θεσμικών οργάνων, φαίνεται ότι η έκθεση αυτή μάλλον θα είναι απλή. Πρώτον, η Επιτροπή Εξωτερικών και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου μας έθεσαν υπόψη κάποια προβλήματα σε σχέση με το άρθρο 90 της Διεθνής Συνθήκης και τη συμφωνία που δίνουμε εμείς, τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου δηλαδή. Και αυτό όμως θα πρέπει να μπει σε ξεχωριστή έκθεση. Εδώ είμαστε ε, στο άρθρο 81 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Επανειλημμένα το έχουμε συζητήσει. Ε, αυτό το θέμα της σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου έχει τύχει διαφορετικής ε, ερμηνείας ε, σε διάφορες επιτροπές όταν πρόκειται για ψηφίσματα, για διάμεσες εκθέσεις, για τροπολογίες και ιδιαίτερα ε, την ίδια την ψηφοφορία. Έτσι, αυτά συνδέονται με διάφορα προβλήματα και με έλλειψη συνοχής τελικά όταν χρησιμοποιείται αυτή η διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το θέμα για μένα το βασικότερο είναι να το διορθώσουμε αυτό και να έχουμε μια ενιαία συνεκτική στάση απέναντι όταν δίνουμε την έγκρισή μας, να σεβόμαστε και το πνεύμα της συνθήκης πάντα, αλλά και τις εξουσίες και τις προνομίες του Κοινοβουλίου. Διότι όταν μπήκε αυτή η διαδικασία έγκρισης, που παλαιότερα ήταν γνωστή ως διαδικασία ε, σύμφωνης γνώμης, ήταν λίγο σαν ένα πυρηνικό όπλο που μπορείς να πεις ναι ή όχι τελικά. Αλλά εμεί είχαμε υπόψη μα μια διαδικασία έτσι πιο διαπραγματευτική για να καταλήξουμε στη συναπόφαση. Ε, και πώς ενισχυθούν οι εξουσίες και τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά όχι με τρόπο που να προσφέρεται για να προσφύγει κανείς στα δικαστήρια. Ιδιαίτερα. Όταν βάζουμε πολλές ε, δικαιολογίες ε, ή επιπλέον όρους ε, για την, στην υπερψήφισή μας, όταν συνδέεται με κάποια αιρεσιμότητα. Λοιπόν, για την απόφαση την ίδια θα πρέπει να είναι απλή, να περιλαμβάνει αιτιολογικές αναφορές, αλλά όχι αιτιολογικές σκέψεις και τροπολογίες, τροπολογίες μόνο σε περίπτωση που δεν συμφωνεί ο συγκητή, δηλαδή να μην βάζουμε όρου στην απόφαση, να είναι σαφές ναι ή όχι. Η, η έγκρισή μας, η, τα υπόλοιπα, μάλλον μη νομοθετικό ψήφισμα θα πρέπει να είναι, που να επισυνάπτεται ε, στην απόφαση. Έχουμε κάποια προβλήματα με καθυστερήσει στην έγκριση, γι' αυτό έχω βάλει την αντίστοιχη παράγραφο για την αρμόδια επιτροπή και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζει ε, τις ε, ολιγορίες και σε σχέση με τη διάσκεψη των πρόεδρων. Τώρα, η σύσταση αυτή καθ' αυτή και η ίδια η ψηφοφορία, γιατί στην Ολομέλεια πολλές φορές υπάρχει σύγχυση. Τι ψηφίζουμε, τη σύσταση ή την ίδια την έγκριση. Τι γίνεται αν είναι αρνητική η σύσταση. Πώς θα γίνει η ψηφοφορία και, και είναι και αρνητική καταψηφιστή. Ε, πώς μπορεί να θεωρηθεί αυτό θετική απόφαση, ιδιαίτερα μετά την ιστορία με την άκτα. Λοιπόν, η λύση ποια να είναι, να είναι άλλο πράγμα η σύσταση, αλλά ψηφίζουμε για την έγκριση, μόνο τη δίνουμε ή την αρνούμαστε, ναι ή όχι. Αυτό είναι για να μην ε, έχουμε... Ε, ψύχηση. Μόνο για την έγκριση ψηφίζουμε ανεξαρτήτως της εγκρίσεως της αρμόδιας επιτροπής, αν εγκρίνει η έγκριση απόρριψη. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη πλειοψηφία ε, θεωρείται ότι δεν εγκρίνεται η πρόταση. Αυτό ε, και νομίζω είναι αρκετά σαφές. Ε, η σύσταση είναι αυτή που είναι. Τι να κάνουμε, δεν είναι δεσμευτική. Είναι κάτι που προτείνει η Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Όταν ψηφίζουμε όμως, ψηφίζουμε επί της έγκρισης αν θα τη δώσουμε ή αν θα την αγκριθούμε και να αποφεύγονται όλες οι συγχύσεις και τα προβλήματα. Και ένα τελευταίο είναι οι ανδιάμεσες εκθέσεις. Το συζητήσαμε και με τους κοιόδης ηγητήρες και μέλη της Επιτροπής Προπολογισμών και μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Οι ενδιάμεσες εκθέσεις είναι σημαντικές, μεν. Οπότε το εγκρίνουμε και αυτό ως ε, έτοιμα. Λοιπόν, αν γίνει αυτή η διευκρίνηση που προτείνω, νομίζω τελικά θα επέλθει και σαφήνεια αλλά και δυνατότητα χρήσης με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα με ενιαίο τρόπο σε όλες τις επιτροπές, έτσι, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και τις για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και με χαρά και προσοχή να ακούσω τα σχόλιά σας. Gualtieri. Συγχαίρω τον Ραφάλ για την εξαιρετική του εργασία. Πρέπει να πω ότι παρουσιάζει μια λογική λύση, αλλά έχω μια αμφιβολία Αλλά είναι απλά αμφιβολία και όχι ακριβώς τροπολογία. Έχω μια αμφιβολία για το κατά πόσο αυτή η λύση θα επικαλύψει την εργασία της Επιτροπής με την εργασία της Ολομέλειας. Γιατί αν η ψηφοφορία στην Ολομέλεια γίνεται χωρίς να λαμβάνει de facto να βάνετε μάλλον de facto υπόψη, γιατί δεν είναι ψήφο της ψηφοφορία τη επιτροπή είναι μια άλλη ψηφοφορία. Βέβαια, αυτό δεν θα είναι μετά από πρόταση της Επιτροπής μας, αλλά σημαίνει πως ένα, μια, ψηφ, μια, αρνητική ψήφος θα γίνει ε, θετική, γιατί θα πρέπει να γίνει μια νέα ψηφοφορία, γιατί η πλειοψηφία μπορεί να είναι διαφορετική αλλά de facto δεν αλλάζει κάτι από αυτά που λες εσύ. Ίσως μόνο το γεγονός ότι εσύ πρέπει να κάνεις μια δεύτερη ψηφοφορία. Ε, μόνος μου φόβος είναι δηλαδή ότι μπορεί κανείς να πει ότι σε αυτή την περίπτωση γιατί να μην πάμε κατευθείαν στην Ολομέλεια που είναι, αφού είναι απλά μία σύσταση. Δεν είναι έκθεση, αλλά δεν είμαι και βέβαιος πρέπει να σας πω. Είναι απλώς μια αμφιβολία. Και φυσικά έχει σημασία και η δυνατότητα να υποβάλει κανείς ένα ψήφισμα Συμφωνώ ότι δεν είναι σωστό να βάλει κανείς μαζί επιχειρηματολογία στο ναι ή στο όχι. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ξεχωριστή έκθεση που θα αναλύει και θα εξηγεί τους λόγους χωρίς να προκαταβάλει την ψήφο. Νομίζω πως de facto αυτή η λύση θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο από ό,τι μπορούμε τώρα, αλλά έχει νόημα να μην, είναι, να μην καταστεί υποχρεωτικό, αν και δεν μου αρέσει ακριβώς η διατύπωση ότι το έχω δώσει στα Ιταλικά, αν περιπτώσει. Δεν μου αρέσει πολύ η διατύπωση. Ο κύριος Ντάφ. Νομίζω πως στην παράγραφο 2 το προτινόμενο άρθρο 81 του κανονισμού ε, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το πολιτικό ψήφισμα, αυτό δεν μπορεί να προκαταβάλει την απόφαση που πρέπει να λάβει το Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι απαραίτητο. Στην παράγραφο 3, μια ερώτηση. Η διάσκεψη των Προέδρων αναλαμβάνει το θέμα τη απουσία σύστασης από την Επιτροπή μας και βάζει το θέμα στην, ολομέλεια της, στην ε, ημερήσια διάταξη με της Ολομέλειας. Όμως η διάσκεψη των Προέδρων επικρατεί της, των προνομίων της Επιτροπής και υποβάλλει δική της σύσταση ή όχι, γιατί αυτό δεν είναι σαφές από τη διατύπωση που έχουμε εδώ. Για ποιο λόγο ακριβώς θα πάει η απόφαση στην Ολομέλεια. είναι για τη συγκατάθεση ή για ουδέτερη προσέγγιση στην Ολομέλεια. Νομίζω πως πρέπει να είμαστε σαφείς και γι' αυτό. Θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε περαιτέρω πριν να ψηφίσουμε. Θα έχουμε άλλη ευκαιρία για συζήτηση στην Επιτροπή μας. Oh, Αυτό το ερώτηση απευθύνεται στον εισηγητή μάλλον. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να ζητά το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον Ραφάλ. Εγώ θα αρχίσω από το τέλος. Νομίζω πως ε, το καλύτερο είναι, δεδομένου ότι δεν είναι και πολλοί που ενδιαφέρονται εδώ, καλύτερα ε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάτσουμε με τους ε, σκιώδεις να συζητήσουμε και να δούμε γιατί βασικά έχουμε να μιλήσουμε για κάποιες ερωτήσεις, κάποια θέματα τα οποία πρέπει κάπως να τα σκεφτούμε περισσότερο. Αρχική μου αντίδραση είναι όταν πρόκειται για τη σύσταση. Η μεγάλη σύγχυση ήταν αν είναι σύσταση, αν είναι τελική ψήφος για συγκατάθεση κτλ. Και δεν ήταν, ε, αυτό το είδαμε σαφώς με την άκτα, όπου αντιστράφηκε ολόκληρο το δόγμα και επί τα άλλες επιτροπές ε, το χειρίζονταν τελείως διαφορετικά. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, αλλά αν έχουμε μια σύσταση πολιτικής φύσης από τη μια δεδομένη επιτροπή μαζί με ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα, νομίζω πως είναι απόλυτα σαφές πως αυτό θα καθορίσει τη διαδικασία, αλλά στο τέλος θα φτάνει στην Ολομέλεια για να αποφευχθεί η σύγχυση θα πρέπει να είναι μια ψήφος ναι ή όχι. Καταρχήν, με το, σύμφωνα με το πνεύμα, τηρείται έτσι το πνεύμα της συνθήκης και έπειτα ε, λύνεται και αυτό το πρόβλημα τι θα γίνει αν έχουμε ναι για όχι ή όχι για το ναι και όλα αυτά. Ξέρω, συμφωνώ πως είναι ριζική λύση, αλλά ε, νομίζω πως είναι και πιο ξεκάθαρη. Τώρα, όπως λέει και ο Άντρου, για το, στην παράγραφο 2 μπορούμε να το αποσαφενήσουμε ότι πρέπει να είμαστε εκεί απόλυτα βέβαιοι πως δεν υπάρχει σύγχυση και εδώ, αλλά εγώ νόμιζα πως ήταν σαφές αυτό που πρότεινα. Τώρα, όσον αφορά την διάσκεψη των Προέδρων, δεν, υποκαθιστά, δεν αντικαθιστά μάλλον την Επιτροπή, αλλά αν δεν γίνεται κάτι στην Επιτροπή, που έχει γίνει πολλές φορές, χωρίς σύσταση, το βάζει στην Ολομέλεια. Δηλαδή, δίνει την τελική ψηφοφορία η Ολομέλεια χωρίς σύσταση αλλά μπορούμε και αυτό να το συζητήσουμε. Αυτό ήταν ε, ένα θέμα που προέκυψε στα τελευταία στάδια της συζήτησης. Τι κάνουμε δηλαδή με τις ε, υπερβολικές καθυστερήσεις. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε για να μην ε, υιοθετήσουμε λύσεις που να είναι αντιπαραγωγικές. Όπως είπα, το συζητήσουμε με τους σκιώδεις, ώστε να μπορούμε μετά όντως να προχωρήσουμε και έπειτα και μετά να ενημερώσουμε τους εισηγητές. Να, τους, τους συντονιστές μας, συγχωρείτε, να, συνεχίσει να προχωρήσει το θέμα. Ο κύριος Νταφ, εντάξει το εκτιμώ αυτό που λες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην ε, ευνοχήσουμε κατά λάθο τις επιτροπές. Να ρωτήσω τον εισηγητή αν θεωρεί λοιπόν σωστό να ορίσουμε με ημερομηνία για την υποβολή ε, τροπολογιών. Μήπως είναι πρόημο? 13 Ιουνίου. Ναι, εγώ νομίζω πως μπορούμε να ορίσουμε προθεσμία. Εμείς θα κάτσουμε παρέα, θα ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα και αν συμφωνήσουμε εντάξει, αν όχι θα υποβάλουμε τροπολογίες και πάμε αμέσω σε συμβιβαστικές. Δεν είναι τόσο, τόσο αντιφατικό το θέμα, ώστε να χρειάζεται περαιτέρω καθυστέρηση. Μάλιστα. 15 Ιουνίου να ορίσουμε λοιπόν προθεσμία. Ναι. Yeah. Όχι, όχι, εντάξει. Αρκεί, αρκεί. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε την εξέταση τη ημερήσια της ε, Τέλος της συνεδρίασης. Χαίρετε.